Hello, good morning. Welcome to all the petitioners. Let's... Καλημέρα, λέει πρώτα. Θα ε, μιλώ στα ισπανικά. Ξεκινούμε. Πρώτα-πρώτα με το σημείο 19 της ημερησίας διατάξεως που είναι η αναφορά 63 κάθετος του 17 του Ιβάιλο Ήλιεφ, βουλγαρικής ηθαγένειας, με 50 υπογραφές για καζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις διαδικασίες εντολών πληρωμής στη Βουλγαρία. Στη συνέχεια, 408 του 17 της Ντεσισλάβα Φιλίποβα, βουλγαρικής ηθαγένειας και άλλες 4.248 υπογραφές για το άρθρο 417 της πολιτικής δικονομίας για παραβίαση δικαιωμάτων των καταναλωτών η 838 του 17 της Βιολέτα Γκοσποντίνοβα, βουλγαρικής ηθαγένειας για εντολή πληρωμής σε σχέση με ενυπόθηκο δάνειο. Επίσης, 514 του 18 του Ιβάιλο Ήλιεφ, βουλγαρικής ηθαγένειας, για διαφθορά δικαστηρίων της Βουλγαρίας και παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη. 606 του 18 της Μιλένα Δημητρόβα βουλγαρικής Σταγένεια, για παραβίαση της οδηγίας 93 κάθετο 13 της Ευρωπαϊκή Ένωση και διαφορά με τράπεζα για στεγαστικό δάνειο. 609 του 2018 της Τσέσκα Χατζηγεωργιέβα, βουλγαρικής σταγένεια, για παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και έλλειψη πρόσβαση σε δικαστήριο. Η 720 του 18 της Βιολέτα Γκοσποντίνοβα, Βουλγαρική ηθαγενεία για απάτη και διαφθορά όσον αφορά την αφαίρεση περιουσία από τράπεζε και δικαστικού επιμελητέ 810 του 18 από κάποιον βούλγαρο πολίτη για την νομιμότητα του άρθρου 417 του Κώδικα Πολιτικής δικονομία για παραβίαση δικαιωμάτων των καταναλωτών σχετικά με εντολές πληρωμής 1045 του 18 από βούλγαρο πολίτη συν άλλες 180 υπογραφές για ασυμβατότητα εντάλματος προσφυγής και έφεσης της ε, πολιτικής δικονομίας. 1193 του 18 από κάποιον βούλγαρο πολίτη από την Ένωση Θυμάτων Διωτικών Δικαστικών Επιμελητών για την Αλληλεγγύη προς τα θύματα ιδιωτικών φορέων επιβολής νόμου και δικαστικού συστήματος 36 του 19 του Δημήτρη Παναγιώτοφ, βουλγαρικής Ιθαγένειας. Από πλευρά τη Ένωση Θυμάτων Ιδιωτικών Δικαστικών Επιμελητών και Δικαστικού Συστήματο, ελεγγύη ε, για διαφθορά και παραβίαση δικαιωμάτων σε δίκαιη δίκη. 37 ε, του 19, Μαριάν Νέλιαβα, ε, Βουλγάρα, σχετικά με παραβίαση του, δικαίου, του δικαίου της Βουλγαρίας. από τη Βουλγαρία για εντολές πληρωμής 40 του 19 από κάποιον ε, βούλγαρο πολίτη σχετικά με τη μη συμμόρφωση από πλευράς βουλγαρικής νομοθεσίας προς τον κανονισμό 1896 του 6 για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής και 51 του 19 της Βασιλιέβα ε, Βουλγάρα σχετικά με την παραβίαση της οδηγίας 93 13 για καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων με καταναλωτές από πλευράς της Βουλγαρίας. Και η 102 του 19 από κάποιο βούλγαρο πολίτη για διαφορά σε σχέση με ενυπόθηκο δάνειο. Έχουμε πολλούς ε, αναφέροντες, οπότε θα πρέπει να καθορίσουμε τι χρόνο έχει ο καθένας στη διάθεσή του και επίσης να γνωρίζετε με ποια σειρά θα μιλήσετε πρώτα-πρώτα. Ο κύριος Ιβάιλο Ήλιο θα μιλήσει πρώτος που μας είπε ότι επίσης έχει να προβάλλει και κάποιο βίντεο. Άρα με το βίντεο έχετε 5 λεπτά. Στη συνέχεια η κυρία Φιλιππόβα Ντεσισλάβα 3 λεπτά. Μετά ο κύριος Σπάσοφ 3 λεπτά. Μετά η κυρία Δημητρόβα 3 λεπτά. Κυρία Σφετλάνα Μιλάνοβα, επίσης, τρία λεπτά. Ο κύριος Νικολάη Πότσεφ, τρία λεπτά. Και στη συνέχεια, πέντε λεπτά, που πρόκειται να κατανείμουμε σε τρεις. Φαβένα Στοντούροφ, Νικολάη Ντασκαλόφ και Νικολάη Κόλεφ. Αυτοί οι τρεις έχουν και οι τρεις πέντε λεπτά. Μετά η κυρία Νατρία Μπράτσεβα έχει τρία λεπτά και ο κύριος Βλάντισταβ Γιάννεφ τρία λεπτά. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση να αρχίσουμε με την ομιλία του κυρίου Ιβάιλο Ήλιεφ. Σας ευχαριστώ και όλοι καλώς ορίσατε από τη Βουλγαρία. Ε, κυρίες και κύριοι, μέλη της Επιτροπής Αναφορών, βλέπετε Όλοι εμείς, όλοι οι αναφέροντες έχουμε έρθει εδώ ενώπιό σας ε, γιατί για μας ε, εδώ είναι ε, η τελευταία λύση. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών θα μας βοηθήσει. και ότι θα διερευνηθούν ε, τα γεγονότα σωστά στην ε, Επιτροπή σας. Ελπίζουμε σε δίκαιη μεταχείριση, ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα λάβει υπόψη της για να ε, υπάρξει κατάλληλη συνεργασία προκειμένου να γίνει ο έλεγχος ε, των γεγονότων. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο πολίτες της Βουλγαρίας, αλλά και πολίτες άλλων χωρών. Είναι σημαντικό να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία επιπαραβάση για τη Βουλγαρία. Το 2016 ο εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, μια μονάδα που διερευνά τη διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο εξέτασε 12 από αυτές τις υποθέσεις μου και πραγματικά βρήκε ότι υπήρξε κατάφορη παράβαση διότι οι δικαστές δεν εξέδιδαν δίκαιες αποφάσεις, δεν υπήρχε πράξη εκτέλεσης η οποία να είναι ε, σωστά συντεταγμένη, ούτε και η επίδοσή τους γινόταν σωστά. Υπήρχε γενικώ ε, μια μεγάλη παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Καθώς καταρχάς οι δανειολήπτες θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Η υπόθεση που εκπροσωπώ είναι η υπόθεση παράνομης απαλωτρίασης κάποιων, ε, κάποιων πάγιων στοιχείων μου. Μάλιστα, ο δικαστικός επιμελητής ε, δεν έδρασε σωστά κομμάτι της ιδιοκτησίας μου, καταστράφηκε, ακόμη και αν δεν ήταν δική μου καθαρά περιουσία, αλλά ανήκε και σε κάποιον άλλον. Ε, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε, δεν ελήφθη κάποια δράση από τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου των ε, δικαστικών επιμελητών στη Βουλγαρία και όλοι θεώρησαν αυτό το συμβάν ότι ήταν κάτι ασήμαντο. Ε, όλα τα ακίνητά μου χρειάστηκε να απαλωτριωθούν σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές αγοράς. Όλα είναι μέσα σε, στο σκοτάδι. Είναι μια, ένα σκοτεινό δωμάτιο που περιλαμβάνει πάνω από 200.000 ε, υποθέσεις παράνομες απαλωτρίωσης ή αντίστοιχων ε, πράξεων που θεωρούνται ότι έχουν κλείσει. Οι ιδιώτες δικαστικοί επιμελητές έχουν επίσης τα έγγραφα στην κατοχή τους έγγραφα για μισό εκατομμύριο πολίτες. Εμείς φυσικά απευθυνθήκαμε σε όλη την ιεραρχία, κανείς όμως ε, δεν ανέλαβε δράση. Γι' αυτό ερχόμαστε σε εσά. Αυτή η εγκληματική πρακτική πρέπει να σταματήσει. Απευθυνθήκαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης, όμως μας είπε πως όλα όσα κάνουμε απλώς δυσφημούν τη Βουλγαρία. Αυτό είναι ε, κάτι σαν απειλή για την οργάνωση και τις δραστηριότητές μας. Υπάρχει διαφθορά στο σύστημα, δεν υπάρχει ανεξαρτησία, δεν υπάρχει τυχαία κατανομή των υποθέσεων. Κυρίες και κύριοι, ε, βασιζόμαστε σε εσά, ε, στην συνεργασία σας, στη βοήθειά σας. Ελπίζουμε να αλλάξει η κατάσταση στη Βουλγαρία, γιατί ε, πραγματικά όλοι εξαρτώμαστε από τους δικαστικούς επιμελητές και σας ευχαριστώ. Πολύ. Σας ευχαριστούμε επίσης που κουτήσατε το χρονικό όριο και τώρα κυρία Μπρισίλαβα. Δεσίσλαβα Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ονομάζομαι Φιλίππο Βαντεσίσλαβο. Και βρίσκομαι εδώ μαζί με τους άλλους αναφέροντες και θα ήθελα να σας πω ότι η αποστολή μας είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και το, τη λύση που δοθεί όταν έχουν παραβιάσει. Το 2014 είχαμε ε, ε, κάνει την αναφορά και ήρθαμε σε επαφή ε, με την Επιτροπή πρώτα-πρώτα και παρουσιάσαμε κάποια πραγματικά περιστατικά και είπαμε ότι η βουλευτική νομοθεσία παραβιάζει την οδηγία 93 του 2013 μια που επιτρέπει ένα σωρό ρήτρες να χρησιμοποιούνται κατά των καταναλωτών. Επίσης, ε, η βουλευτική νομοθεσία επιτρέπει στο να υπάρχουν διάφορες παγίδες στις συμβάσεις. Επίσης, χρησιμοποιούνται κάποιες συνοπτικές διαδικασίες κατά των καταναλωτών, οι οποίοι έχουν λάβει κάποια δάνεια. Οπότε παρακολουθείτε στενά και υποπτεύετε από αυτή την πλευρά η Βουλγαρία και ξεκίνησαν κάποιες ε, διαδικασίες κατά της χώρας. Παρ' όλα αυτά, εμείς συνεχίζουμε αυτή μας την αναφορά, διότι παρά τη διαδικασία παραδιάση κατά της Βουλγαρίας, οι Βούλγαροι νομοθέτες συνεχίζουν, συνεχίζουν την προηγούμενη γραμμή τους. Και επίσης έχουν και κάποια νομοσχέδια τα οποία επεξεργάζονται και έχουν κατευθεί στο Κοινοβούλιο. Τα οποία νομοσχέδια ε, αποτελούν αντικείμενο στο οποίο έχω και εγώ ασχολήθει και αφορά πάλι κάποιους ε, κατά των οποίων τελικά επιβλήθηκαν μέτρα όπως πάγωμα των περισσοικών των στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών. Δηλαδή συνεχίζεται αυτού του είδους η τακτική κατά των καταναλωτών. Οι αρχέ τώρα της Βουλγαρίας θα καθυστερήσουν την ε, τροποποίηση των νομοθετημάτων. Αλλά τελικά θα περάσουν ε, τους νόμους που θέλουν, που είναι κατά των καταναλωτών και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Και να σας πω δύο λόγια. Ε, ε λέει άλλη κυρία, έχουμε το άρθρο 417 στη χώρα. Είναι ένα άρθρο αυτό από την κώδικα ποινική δικονομία. Ε, εσείς μιλάτε από το χρόνο της κυρίας ναι. Και εγώ για την ίδια υπόθεση για την ίδια αναφορά, λέει ο ομιλούσα. Οπότε, βρισκόμαστε εδώ για να σας ζητήσουμε να ε, βοηθήσετε σε σχέση με αυτούς τους νόμους. Έχουν γίνει επομένω κάποιες τροπήσεις της νομοθεσίας. Αυτές έχουν υποβληθεί για έγκριση στο Κοινοβούλιο, αλλά ε, τελικά δεν εξυπηρετούν καθόλου Τελικά αυτή η τροποποίηση του δικαίου ωφελεί τα μονοπόλια στη χώρα. Ούτε κατά όλες αυτές τις διαδικασίες ανταποκρίνονται στα αιτήματά μας, δεν μας δίνουν απαντήσεις σε αυτά που ρωτούμε. Ό,τι έγινε, έγινε από τον διαμεσολαβητή που βρίσκεται σε συνεχή προστρεβή με το Κοινοβουλίο. Άρα λίγα πράγματα έχουν γίνει και οι τροποποίησεις του νόμου δεν βελτιώνουν την θέση του καταναλωτή. Οπότε θα πρέπει να πιέσουμε τις αρχές να δώσουν σχετικές πληροφορίες, αλλά, αλλά σιωπούν οι αρχές. Σβέτοσλαφ Σπάσοφ τώρα. Κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε τρεις αναφορές ε, μέσα σε τρία λεπτά. Να σας εξηγήσω ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Η ιδιοκτησία του αναφέροντος πουλήθηκε της αναφέροντος πουλήθηκε προτού καν να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία εναντίον της. Το βουλγαρικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η σύμβαση πώλησης της ιδιοκτησίας μπορεί ε, να είναι ε, άδικη, με, σύμφωνα με άδικους όρους. Η απόφαση του δικαστηρίου δήλωνε λοιπόν ότι οι όροι του συμβολέου δεν ήταν δίκαιοι και ότι ανεξάρτητα από αυτό έγινε νόμιμα η πώληση της ιδιοκτησίας. Ε, οπότε η αναφέρουσα δεν είχε δικαίωμα σε αποζημίωση. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε εάν το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζεται στη Βουλγαρία και σε τι βαθμό. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, δεν εφαρμόζεται καθόλου. Να σας θυμίσω ότι η σχετική οδηγία δείχνει πως ε, Πολλά προβλήματα αναλύθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχουν βρεθεί λύσεις σε κάποιο βαθμό. Όμως ένα από τα εμένοντα προβλήματα φαίνεται να είναι η αποτελεσματικότητα και η δικαιοσύνη. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εφαρμοστεί σωστά το κοινοτικό δίκαιο από τα κράτη-μέλη δεν βλέπουμε πρόληψη των κακών πρακτικών. Επίσης, οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα είχαν απόλυτο δίκιο. Αν δούμε τη διοικητική πλευρά, όντως όλοι οι κανόνες και οι κανονισμοί εφαρμόστηκαν. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Εμείς ως πολίτες δεν είμαστε προστατευμένοι. Άρα ποιο το νόημα της ύπαρξης κοινοτικού δικαίου. Αυτό το πρόβλημα δεν υφίσταται μόνο στη Βουλγαρία. Θα ακούσετε και άλλους αναφέροντες. Και θα δείτε ότι τελικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αποφασίσει σχετικά με μια υπόθεση στην Πολωνία όπου και πάλι δεν εφαρμόστηκε σωστά το κοινοτικό δίκαιο. Άρα, κάνω έκκληση σε εσά, αναφέρομαι σε εσά ε, για να μπορείτε να έχετε ε, συνέχεια ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της διαδικασίας επί σε τέτοιες υποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μιλένα Δημητρόβα έχει το λόγο. Благодаря. Ευχαριστώ πολύ. Η υπόθεση του πελάτη μου που παρίσταται σήμερα εδώ σχετίζεται με πολλαπλές παραβιάσεις της οδηγίας 93-13 η δίκαιη δίκαιη και η σωστή αποκατάσταση ε, ε, για τον πελάτη μου είναι κάτι που πραγματικά ορίζει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Το πιο σημαντικά πραγματικά περιστατικά είναι τα εξής. Καταρχάς, Η αναφέρουσα για πολύ καιρό ε, πολύ καιρό πριν ε, παραπλανήθηκε και πήρε ένα δάνειο στεγαστικό χωρίς να τη ρωτήσουν ποιος είναι ο μισθός της. Δεν έδωσε λεπτομέρειες στην τράπεζα. Στη συνέχεια, οι δόσεις ε, του δανείου από 346 ευρώ το μήνα πήγαν στα 782 συν μια πληρωμή εφάπαξ 1000 ευρώ ανά έτος. Αυτό στην πράξη σήμαινε ότι έπρεπε να πληρώνει 783 ευρώ το μήνα, αλλά μόνο τα 99 από αυτά πήγαιναν στην ουσία στο δάνειο. Όλα τα υπόλοιπα ήταν για τέλη εξυπηρέτηση του δανείου από την πλευρά της τράπεζας. Αυτά όλα χωρίς να ορίζονται ξεκάθαρα στους όρους του δανείου. Υπήρξε λοιπόν παραπληροφόρηση. Παραπλανήθηκε η πελάτη μου διότι αυτό που της είπε η τράπεζα είναι ότι εφόσον δεν απέδειξε το εισόδημά σου και το είχε όταν έκανε το σύμβαση του δανείου, όμως δεν τη ζήτησαν να το κάνει. Αφού λοιπόν δεν απέδειξε το εισόδημά σου, μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα μέτρα εναντίον σου. Θεωρώ ότι αυτό είναι παραβίαση των δικαιωμάτων της. Επίσης, από την πλευρά του Αγγελέως και της αστυνομίας ε, υπήρξε καταστολή, ε, κατασταλτική δράση εναντίον του γιού της. Όταν αυτή ε, προσπάθησε να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της, όντως το δικαστήριο διαπίστωσε ότι υπήρξε παραπλάνηση, Όμως, ε, οι πρωτόδικες αποφάσεις ε, δεν ήταν σωστές, επομένως έπρεπε στο τέλος να καταβάλει όλα τα ποσά που είχε υποχρεωθεί να πληρώσει ε, στους ανθρώπους αυτούς επειδή την εξαπάτησαν. Παρακαλώ κρατήστε αυτή την αναφορά ανοιχτή και κρατήστε και όλες τις αναφορές ανοιχτές για να μπορούμε να έχουμε σωστά και αποτελεσματικά ένδικα μέσα και δίκαιες δικαστικές διαδικασίες στη Βουλγαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Εσπέλα Μιλανόβα έχει το λόγο, παρακαλώ. Уважаеми дами и господа, от Комисията по петиции Κυρίες και κύριοι, μέλη της, Αναφορών, σας παρουσιάζω την, την υπόθεση της κυρίας Γεωργίεβα, η οποία είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική. Είναι κλασική υπόθεση, ένα άτομο που πήρε δάνειο και στη συνέχεια πουλήθηκε η ιδιοκτησία το ακίνητο. Η συγκεκριμένη πελάτησα ποτέ δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει τα ε, δικαιώματά της ως καταναλώτρια. Δεν μπόρεσε ποτέ να προσφύγει κατά των άδικων όρων της σύμβασης. Κατά την ακρόαση της ε, υπόθεσης συνέβη αυτό, όχι όμως κατά την εκτέλεση. Η Οι δικαστικοί επιμελητές ε, στην ε, ε, Βουλγαρία και γενικά η διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων είναι όλα μέσα στον, σε μια διαδικασία παράνομη και οι πελάτες, οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τα δικαιώματά τους και πολλές φορές ακόμα και όταν πηγαίνουν στο δικαστήριο δεν θεωρείται παραδεκτή η προσφυγή τους. Ε, φαίνεται λοιπόν ότι το σύστημα στη Βουλγαρία έχει απογοητεύσει τους πολίτες, τους καταναλωτές. Δεν φαίνεται να τους προστατεύει και αυτό πιστεύουν και οι καταναλωτές. Φυσικά θέλουμε δίκαιη δίκη, όμως αυτό δεν ισχύει Φυσικά, οι πολίτες της Βουλγαρίας αισθάνονται απογοήτευση. Και αυτός είναι και ο λόγος που είμαστε όλοι σήμερα εδώ. Οι Βουλγαροί πολίτες ε, στρέφονται προς τους βουλγαρικούς θεσμούς, αλλά ε, πάντοτε βλέπουν ότι υπάρχει αμέλεια από την πλευρά τους. Και το σύστημα της Βουλγαρίας μοιάζει με ένα κλειστό κύκλο που αρνείται να ανοίξει και να εξετάσει οποιαδήποτε προσφυγή των βούλγαρων πολιτών και των εκπροσώπων τους ε, στο δικαστήριο. Να πω ότι κάποιοι από τους ε, δικηγόρους είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι και γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Όμως, τα βουλγαρικά δικαστήρια δεν τα θεωρούν αυτά αρκετά σημαντικά. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το σύστημα των δικαστηρίων στη Βουλγαρία δεν είναι ανεξάρτητο. Δεν μπορεί να εκπληρώσει τη βασική του ε, αρμοδιότητα ως ένας από τους θεσμούς του δικαστικού συστήματος. το σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα να προστατέψει τα δικαιώματα των πολιτών. Εμείς, οι Βούλγαροι, είμαστε επισήμως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να ασκήσουμε τα δικαιώματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται στους άλλους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει μια διαδικασία παρακολούθησης. Από την πλευρά σας, τα τελευταία χρόνια έγιναν κάποιες ε, προσπάθειες, ε, έρευνες και μας βοηθήσατε πολύ. Είμαστε ευγνώμονες γιατί υπήρξε κάποια πρόοδος. Ε, αυτή τη στιγμή οι βουλγαρικοί θεσμοί προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να μιμηθούν ότι υπάρχει μια βελτίωση, αλλά δεν είναι πραγματική βελτίωση και γι' αυτό συνεχίζουμε να προσφεύγουμε σε εσά και να ζητούμε τη δράση. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Νικολάη Μποτσέφ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία που μου δίνεται για να εκπροσωπήσω τον πελάτη μου, να μιλήσω εξ ονόματός του, να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και τους ε, για την εξέταση της αναφοράς του πελάτη μου σε αυτή την συνάντηση σε αυτή την συνεδρίαση, όπου σας παρουσιάζουμε την αναφορά μας για να την εξετάσετε. Μετά την αποδοχή της αναφοράς από την Επιτροπή σας, μετά δηλαδή που έγινε δεκτή για να εξεταστεί από την Επιτροπή σας, έχουν προκύψει κάποιες άλλες περιστάσεις νέες σε σχέση με τις διαδικασίες για την ιδιωτική περιουσία, την ιδιοκτησία του πελάτη μου. Και τον έβγαλαν από την ιδιοκτησία του. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα στην πράξη του πώς υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα στο δικαστικό σύστημα στη Βουλγαρία. Νομίζω ότι συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το άρθρο 417 ε, του κώδικα ποινική δικονομίας. Πολλοί από τους συναδελφούς ήδη το ανέφεραν. Δεν πρόκειται να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού. Όμως ε, η παρατήρηση στέκει πιστεύω. Το ε, δεύτερο μου σχόλιο έχει να κάνει με τον ε, αστικό κώδικα. Και με τις διάφορες πράξεις για τις οποίες μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε προσφυγή ή έφεση, τα δικαστήρια συχνά ε, εκδίδουν ομολογία αντιφατική, διότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο κείμενο νομοθετικό σχετικά με τη λύση μιας σύμβασης λόγω ε, ε, έλλειψης, απουσίας ή αδυναμίας πιστωτή. Το άρθρο 743 Ε, δεν επιτρέπει στον πελάτη μου να υποβάλει προσφυγή, να προσφύγει ενάντια στα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί σε βάρος του. Άρα τυπικά την υπόθεση χρειάστηκε να εξετάσει το δικαστήριο. Όμως δεν μπόρεσε το δικαστήριο να εξετάσει επί της ουσίας την υπόθεση. Είναι δηλαδή ένας διαδικαστικός κανόνας, ο οποίος στην πράξη κατάφορα περιορίζει την πρόσβαση του πολίτη στο δικαστικό σύστημα. Γιατί το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει μόνο το τυπικό της υπόθεσης και όχι την ουσία. Και αυτό αποβαίνει σε βάρος των πολιτών. Ένα άλλο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω έχει να κάνει με τους ιδιώτες δικαστικούς επιμελητές. Το καθεστώς των οποίων θεωρείται στην πράξη ισότιμο με αυτό των κρατικών αρχών από τη μία και από την άλλη όμως δεν έχουν διοικητική ευθύνη. Δεν έχουν υποχρέωση ε, να απολογηθούν σε σχέση με τις πράξεις τους ή τις παραλήψεις τους κατά την άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων. Υπάρχει λοιπόν η αστική ευθύνη Μπορεί όμως να ξεκινήσουν τέτοιες διαδικασίες περιαστικής ευθύνης αλλά είναι πάρα πολύ περίπλοκες και επαχθείς για τον μέσο βουλγαριό πολίτη. Στοιχίζουν πάρα πολύ, πρέπει να προσλάβουν δικηγόρο για να στραφούν εναντίον του ιδιώτη δικαστικού επιμελητή. Δεν είναι σωστός το τρόπος αυτός, δεν προασπιζόμαστε έτσι τα δικαιώματα των πολιτών και δεν ε, εφαρμόζουμε με δίκαιο τρόπο τον νόμο. Και γι' αυτό θα πρέπει να λυθεί οριστικά αυτό το πρόβλημα. Το κράτος αγνοεί το πρόβλημα ενώ είναι συστηματικό. Και γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Γι' αυτό προσφεύγουμε σε εσά. Και γι' αυτό βλέπετε τόσες πολλές αναφορές και αναφέροντες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σάμπεν Ασταρούντοφ, ο κύριος Νικολάη Ντάσκαλοφ και ο κύριος Νικολάη Τολέφ. Και οι τρεις θα έχουν πέντε λεπτά από κοινού. Παρακαλώ. Ο κύριος Νικολάη Δασκαλόφ. Είμαι βούλγαρος δικηγόρος. Του, εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του μεγάλου ιδιωτικού κεφαλαίου με τον κώδικα πολιτικής οικονομίας έτσι όπως έχει οθετηθεί στη Βουλγαρία. Πολύ μικρές αλλαγές ίσονος ε, σημασίας έχουν γίνει μετά από τις παρενέσεις της Επιτροπής. Και το άρθρο 417,8 του αστικού κώδικα αποφεύθηκε τελευταία στιγμή, το οποίο ήταν κατάφορα ντροπιαστικό για τη βουλγαρική δικαιοσύνη. Υποτίθεται ότι με αυτό οι τράπεζες μπορούν να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση με βάση μόνο δικά τους έγγραφα, ιδιωτικά δηλαδή των τραπεζών, χωρίς κανένα μία άλλη απόδειξη ε, από άλλη πηγή. Ε, καταστράφηκαν επιχειρήσεις, καταστράφηκαν πολίτες. Και όλα αυτά έχουν συμβάλει στην καταβαράθρωση των οικονομικών του κράτους και όλο αυτό οφείλεται στην αδιφαγία ορισμένων ομίλων, επιχειρηματικών, μεγάλων ομίλων στην κοινωνία μας. Φανταστείτε σήμερα να μαθαίνετε ότι έχουν θεσμευτεί οι τραπεζικοί σας λογαριασμοί και ότι η μοναδική σας κατοικία έχει βγει στο σφυρί με τη μισή τιμή και δεν μπορείτε να αντιδράσετε, ε, ακόμα και αν έχετε εύλογες αντιρρήσεις και ενστάσεις. Στη Βουλγαρία αυτή η κατάσταση επικρατεί. οι ιδιώτες, οι δικαστικοί επιμελητές δεν επιδίδουν αυτές τις ε, κοινοποιήσεις. Στρέφονται εναντίον ε, τυφλών ή αναπήρων ή ε, ατόμων πολύ προχωρημένης ηλικίας. Δεν μπορεί κανείς να σταματήσει αυτή την εντολή, ακόμα και αν υπάρχουν διαδικασίες ερευνητικές ανεξελίξεις στην όλαφη στις Εθνικές Αρχές κατά της διαφθοράς. Διατάσσεται άμεση εκτέλεση του κατασχετηρίου και πνίγεται ουσιαστικά στα χρέη ο φιλέτη. Για τα μάτια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα πάντα είναι δυνατά στη Βουλγαρία. Όταν γίνεται συζήτηση για το κώδικα πολιτική δικονομία και τα δικαιώματα των καταναλωτών, αυτό είναι καλό. Ελπίζω όμω να μην χάσουμε από μπροστά μα το τεράστιο πρόβλημα των μεγαθυρίων, των τραπεζών, τα οποία, οι οποίε τράπεζε έχουν μετατραπεί σε τέρατα, σε θηρία, τα οποία καταδικάζουν τα άτομα καταδικάζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ρουφούν σαν βαμπύρ ε, το αίμα ε, από τη σφίζουσα οικονομία της χώρας μας. Νομίζω ότι ε, έχουν επιληθεί διάφορα θέματα με τις προτάσεις που έχουν υιοθετηθεί. Όμως, γίνεται κατάχρηση του νόμου και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους ιδιώτες δικαστικούς επιμελητές. Είναι ιδιώτες, δεν τους ελέγχει κανείς. Γίνεται καταστρατήγηση του άρθρου 181 ε, του συντάγματος. Ε, χρησιμοποιούνται οι τράπεζες για να εκαθαριστεί ο εμπορικός ανταγωνισμός και να υπάρξουν ολιγοπόλια δεν περιμένουμε ότι θα επιληθεί το θέμα με τις επικείμενες τροπολογίες. Η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των βουλγαρικών αρχών δεν μας ε, δίνουν καμία ελπίδα. Έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για άλλο έναν συμβασμό που είναι έτοιμη η Ευρώπη να κάνει ε, για να εξυπηρετήσει τα διάφορα πολιτικά λόμπι. Ε, ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ζητήσει από την Επιτροπή να αναλάβει τις ευθύνες της και από το βουλγαρικό κράτος, γιατί έλυσαν με ατελή τρόπο ό, όλα αυτά τα προβλήματα και δημιούργησαν νέα τα οποία ε, βασανίζουν τους αναφέροντες σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι, λέγομαι του Στουντούροφ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών γιατί μου έδωσε το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τίμερμαντς, τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Και θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα της Όλαφ που ασχολήθηκε με το φάκελο 1079 του 2017 την διερεύνηση της C-Bank που είναι θηγατρική της βελγικής ΚΑΜΠΕΣΕ. Και για να, θέλω να σας εξηγήσω γιατί υπέβαλα την αναφορά. Το 1987 ε, ένας ε, μια επιχείρηση τηλεγραφημάτων έστειλε ένα τηλεγράφημα σε διάφορα προξενία και είπε ότι είναι 21 Ιουνίου, οι χριστιανοί στην Κοαπάρνα σφαγιάζονται και αν δεν υπάρξει βοήθεια που να σταλεί μέχρι αύριο θα σκοτωθούν όλοι. Και παρακαλώ προωθήστε αυτό το τηλεγράφημα σε όλους μας τους πρέσβεις. Ήταν συγγενής μου λοιπόν αυτός ο χειριστής, ο τηλεγραφητής και χάρη στην άμεση ανταπόκριση ε, διπλωματών Ευρωπαίων. Πάνω από 5.000 Βούλγαροι από αυτή την περιοχή διασώθηκαν από το θάνατο και την καταστροφή. Προσφεύγω λοιπόν σε εσά ε, σήμερα και σας ζητώ να αναλάβετε έγκαιρη, γρήγορη δράση για να σταματήσετε αυτή τη δεκαετή λαϊλασία που έχουν υποστεί οι Βούλγαροι πολίτες σε καιρό ειρήνης. Ελπίζω ότι η διαδικασία επί παραβάση δεν θα προκαλέσει οικονομικές κυρώσεις στη Βουλγαρία γιατί έτσι θα αυξηθεί μόνο το βασανισμό, το βανεστήριο, το άχθος, το βάρος που φέρουν οι πολίτες. Πρέπει να απολογηθούν οι νομοθέτες οι οποίοι ευθύνονται για την τρέχουσα κατάσταση. Περιμένω γρήγορα έγκαιρη δράση, αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Μην ξεχνάτε τα τρίτα μέρη που έχουν ε, υποστεί τεράστια ζημιά ως καταναλωτές σε αυτό το πλαίσιο της ε, ε, εσφαλμένης και φαύλης εντολής πληρωμής και των διαδικασιών. Η οικογένειά μου, εμείς έχουμε υποστεί αυτή τη ζημία και η η απάντηση που έλαβα πριν από λίγες μέρες, την απάντηση του Υφυπουργού Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση και πρέπει να σας πω ότι συνοψίζεται στο εξής. Είναι μια άνευ προηγουμένου ομολογία και θέλω να σας διαβάσω και να παραθέσω τι λέει ο Υφυπουργό. Και παραθέτω, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας στη Βουλγαρία δεν περιλαμβάνει τους αντίστοιχους κανόνες που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τέλος της παράθεσης. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου. Είναι ξεκάθαρη ομολογία αυτό. Και αποδεικνύει ότι έχουμε δίκιο. Και καλώς υποβάλλουμε αυτή την αναφορά. Όλες οι αναφορές των βουλγαρών πολιτών είναι πολύ σωστά τεκμηριωμένες. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρέπει να σας αναφέρω για το ότι ο κώδικας πολιτικής δικονομίας είναι προκειμένου αφήνει το περιθώριο τους ώστε να έχουμε αυτή τη συμμορία των τραπεζών, των δικαστικών ε, κλητήρων, ε, των εισαγγελέων, των δικαστών. Ε, αυτό είναι φανερό. Ξέρετε, είχαμε ένα σωρό δίκες με αφορμή αυτές τις διαταγές πληρώμησης. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρο, και τώρα η κυρία Μαρία Αμπράσεβα. Κυρίε και κύριοι, Επιζητώ με τη βοήθειά σας. Να δούμε τι θα γίνει με αυτές όλες τις ε, δίκες για τις τεταγές πληρωμής. Βουλγαροί, γενικότερα Ευρωπαίοι, αλλά ακόμα και πολίτες τρίτων χωρών που ζουν στην χώρα μας, στην πράξη, στερούνται του δικαιώματος προστασίας τους ως καταναλωτές. Άρα δεν εφαρμόζεται η οδηγία 93-13. Η προστασία αυτή συντρέχει ακόμα και αν δεν έχει κάνει τη σχετική καταγγελία ο καταναλωτέ. Πολλέ φορέ πάντω στη χώρα μα. οι τράπεζε επικαλούνται το άρθρο 417 και ασκούν τι σχετικέ αγωγέ. Είναι δύνατον να περάσει από έλεγχο η σύμβαση γιατί δεν απαιτείται από την τράπεζα να υποβάλει προς έλεγχο το περιεχόμενο των ε, συμβάσεων. Γι' αυτό σας λέω ότι στην πράξη ο νόμος είναι αναποτελεσματικός. Πολύ συχνά οι δικαστές ξεργάζονται με τις ε, ιδιωτικές εταιρείες των ε, δικαστικών επιμελητών. Στη Γαλλία είχαμε παρόμοιες περιπτώσεις όπου είχαν παρέμβαση Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ αυτό δεν έχει συμβεί στην Γαλλία. Πάντω, η εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων γίνεται και κλεισμένα των θηρών. Πολλέ φορέ γίνεται ε, εν κρυπτό ω προ τον οφειλέτη και εκείνο μια ωραία μέρα βλέπει να του έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία, που το έχουν δεσμεύσει τέλο πάντων. Ο φιλέτη δεν μπορεί καν να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και σας λέω ότι είναι προβληματικό αυτό το σύστημα των ε, ιδιωτών δικαστικών κλητήρων. Παρά είναι ισχυρέ οι τράπεζες. Και αυτό περιορίζει τον ανταγωνισμό. Επίσης, αυτό αποτελεί κλοπή της ατομική ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε, κρατήστε ανοιχτές τις αναφορές και συνεχίστε να ασκείτε πίεση στην Βουλγαρία για να μπορέσουν τελικά οι βουλγαρικές αρχές να ευθυναμίσουν την νομοθεσία μας με το κοινοτικό δίκαιο. Πρόκειται για τα δικαιώματα τα οποία έχουμε στους Ευρωπαίοι πολίτες. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα. Το λόγο έχει ο Βλάντισλαβ Γιάννεφ. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, συμφωνώ με όλα όσα είπαν οι άλλοι αναφέροντες που εκπροσωπούν τον λαό μας. Είναι μία τραγωδία. Μας ληστεύουν. Μιλούμε για κάποιες διαδικασίες που έχουν θεσπίσει και που αποτελούν το άκρονάδον της παρανομίας. Πρόκειται για κάποιες διαδικασίες που καταλήγουν στην λίστευση της περιουσίας των ε, Βουλγάρων. Και αυτό μέσα από μια διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. Έχω όλα τα στοιχεία να τα δώσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και έχω αυτά τα στοιχεία από το 2014. Πρόκειται για κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Σε αυτές τις αποφάσεις ματιώνεται η εφαρμογή, ε, εφαρμογή και εκτέλεση κάποιου εντάλματος κάποιης διαταγής πληρωμής. Αυτή η απόφαση ορίζει, καταλήγει στο ότι υπάρχει ασυμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική. τα δικαστήρια στη χώρα δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Επίση έχουμε και κάποια έφεση. Προσφυγή τέλο πάντων και αφορά κατά δίκη βουλγαρου να καταβάλει στην τράπεζα χωρίς να έχει δικαίωμα προσφυγής. ίδιοι δικαστές πρόκυψε ότι έχει πάρει δάνεια από την ίδια τράπεζα, εκείνη που ήταν ο ενάγωνος στην υπόθεση. Και στη συνέχεια κάποια από τα έγγραφα της διαδικασίας είχαν παραποιηθεί και πλαστογραφηθεί. Στη συνέχεια οι ίδιοι δικαστές κατήγγειλε τον αναγόμενο ε, και τελικά όμως η δικαστής εκρίθη ότι είναι ένα δίκο και σύμφωνα με το νότο του πειθαρχικό όργανο ε, εγώ ήμουν ο συνήγορος του συναδέλφου που είχε συρθεί στο δικαστήριο από τη δικαστήνα ε, τώρα έχει αποστερηθεί την άδεια του επαγγέλματος αλλά όλα αυτά σας λέω ότι είναι ε, παράνομα. Με όλα αυτά θέλω να συμπληρώσω αυτά τα οποία ήδη ακούσατε για την παρανομία στην οποία έχουν καταλήξει οι τράπεζες στη Βουλγαρία και έτσι με τέτοια, τέτοιες εντολές πληρώμες κερδίζουν. Πολλοί συνάδελφοι στην χώρα βέβαια δουλεύουν για τις τράπεζες. Επομένως, πρόκειται για διαφθορά στο ανώτατο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής οι πολίτες. Δεν μπορούν με ενδικά μέσα να δικαιώσουν τα δικαιώματα τους, διότι ε, καταστέλλονται ε, και οι ίδιοι οι δικηγόροι που όταν θέλουν να κάνουν ε, το, το λειτουργήμά τους τους απειλούν. Τους απειλούν ότι θα τους αφαιρέσουν τα δικαιώματά τους, την άδεια εργασία τους. Οπότε όλα αυτά είναι πάρα πολύ επιβλαβή για Βουλγάρους και ξένους που στη Βουλγαρία. Είναι φυσικά πολύ κακά για τις ξένες επενδύσεις. Η κυβέρνηση εννοείται ότι δεν σκοπεύει να κάνει τίποτα για αυτή την κατάσταση. Οπότε ε, ελπίζω εσείς κάτι θα κάνετε έγκαιρα και αποτελεσματικά. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους αναφέροντες και τώρα για να αρχίσουμε τον ε, γύρο των παρεμβάσεων και πρώτα, πρώτα ο κύριος Ρόμπερτ Μασιάκ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί αναφέροντες, ε, για τις δηλώσεις σας σήμερα το πρωί, για τις καταθέσεις σας. Φαίνεται ε, ότι έχετε καταθέσει κάποια προβλήματα του βουλγαρικού συστήματος όχι μόνο προς τις διατάξεις αλλά και ως προς τις πρακτικές ε, ιδιωτών όπως είναι οι ιδιώτες δικαστικοί επιμελητές. Αναφέρθηκαν συγκεκριμένες περιπτώσεις πολιτών που έχασαν την περιουσία τους και θεωρούν ότι δεν είχαν μια δίκαιη δίκη. Την ίδια στιγμή είναι σημαντικό επίσης να τονίσουμε ότι ε, οι κανονισμοί στα αστικά ζητήματα, ειδικά ως προς ε, τις εντολές πληρωμής, δεν έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, οι κανόνες αυτοί και η εφαρμογή τους σε μεγάλο βαθμό εμπίπτουν στο εθνικό δίκαιο. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέσα από το δίκαιο της δημιουργήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για διασυνορικές υποθέσεις όπως ο κανονισμός για τις εντολές πληρωμής είναι κάτι διαφορετικό. Η Κομισιόν μπορεί να παρέμβει μόνο στις περιπτώσεις που το κοινοτικό δίκαιο ρυθμίζει συγκεκριμένες πτυχές, κάποιους κανονισμούς ή την ε, εφαρμογή τους, ε, την εφαρμογή κυρίως δικαιωμάτων που προκύπτουν από το κοινοτικό δίκαιο, όπως για παράδειγμα την προστασία των καταναλωτών ε, εναντί ε, των προδιατυπωμένων συμβολέων και των άδικων όρων τους, σύμφωνα με την Οδηγία 9313. Η οδηγία στο χάρτη των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων μιλά για αποτελεσματικά ενδικά μέσα ε, που διασφαλίζουν την προστασία έναντι των άδικων όρων. Σε πάρα πολλές υποθέσεις το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει θεσπίσει αρχές ε, και πρότυπα για σε σχέση με το θέμα αυτό. Επίσης, η καθοδήγηση της 22ης Ιουλίου του 2019 από την Κομισιόν για την οδηγία για τους άδικους όρους καλύπτει αυτή το νόμο με έναν τρόπο ε, ξεκάθαρο. Υπό αυτή την έννοια, οι εθνικοί κανονισμοί δεν θα πρέπει να δυσκολεύουν τους καταναλωτές να βρουν προστασία έναντι ε, κάποιων άδικων όρων, ειδικά όταν μιλάμε για προδιατυπωμένα συμβόλαια. Αυτό σημαίνει ότι τα εθνικά δικαστήρια πρέπει να αξιολογήσουν τη δικαιοσύνη των όρων, ακόμα και αν οι πολίτες δεν έχουν θέσει το θέμα. Γιατί πολλές φορές οι πολίτες δεν γνωρίζουν καν τα δικαιώματά τους. Ε, κάποιες από τις αποφάσεις ε, των δικαστηρίων αφορούν συγκεκριμένα τη διαδικασία εντολής πληρωμής το δίκαιο του καταναλωτή απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες ως προς τις ε, ε, εκδόσεις ε, διαταγής πληρωμής αλλά και για την άμεση εκτέλεσή τους. Έχει ξεκινήσει το 2019 μια διαδικασία επί παραβάση από την Κομισιόν κατά της Βουλγαρίας και αφορά και στο άρθρο του 417 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας που ανέφεραν πολλοί από τους αναφέρονται σήμερα. Το Μάρτι του 2019 η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ενημέρωσε την Κομισιόν ότι είχε καταθέσει νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο για να ενισχύσει τις διαδικαστικές εγγύσεις για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που λάβαμε από τις βουλγαρικές αρχές, Ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή ε, η πρόταση είναι στη δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας και αναμένεται να ε, εγκριθεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2019. Το τελικό, η τελική μορφή των διατάξεων ε, θα εξαρτηθεί βέβαια από την νομοθετική διαδικασία, άρα μόνο στο τελικό στάδιο μπορούμε να αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές βελτιώσεις για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, προτείνεται όταν υπάρχει διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ο καταναλωτής να καταθέτει τους γενικούς όρους του συμβολέου και να μπορεί το δικαστήριο να τους ελέγχει πριν να εκδώσει ε, αυτή τη διαταγή πληρωμής. Επίσης υπάρχουν βελτιώσεις ως προς ε, τα δικαιώματα των πολιτών να αντιταχθούν σε μια τέτοια εντολή. Επίσης οι αρχές της Βουλγαρίας μπορούν να πάρουν επιπλέον μέτρα για να μπορέσουν να διασφαλίσουν καλύτερη συμμόρφωση με τους ε, εθνικούς εθνικούς κανονισμούς. Ας πούμε, ε, πώς ακριβώς δρούν οι δικαστικοί επιμελητές, οι ιδιώτες επιμελητές. Όμως η Κομισιόν δεν έχει στο δικονομικό δίκαιο δικαιοδοσία και δεν μπορεί να εξετάσει όλα αυτά τα θέματα που έθεσαν οι αναφέροντες. Ας πούμε, σε κάποιο βαθμό βλέπουμε ότι υπάρχει παραβίαση του βουλγαρικού δικαίου Επιπλέον η Κομισιόν δεν μπορεί να παρέμβει σε ατομικές υποθέσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιον των βουλγαρικών δικαστηρίων. Η Κομισιόν θα παρακολουθεί στην περαιτέρω πρόεδρο στην Βουλγαρία ως προς τη διαδικασία επιπαραβάση και αν είναι απαραίτητο θα σκεφτεί να λάβει και επιπλέον μέτρα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχουν τα μέλη της Επιτροπής. Ο κύριος Τούδα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πολωνικά. Κυρίες και κύριοι, ο συνάδελφος Ασίμα Κοπούλο ή συνάδελφος μου ζήτησε να την αντικαταστήσω και να παρουσιάσω τη γνωμοδότησή της για τις διάφορες αναφορές για το άρθρο 417 του Βουλγαρικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας σε σχέση με τις διαδικασίες ιδιωτικής εκτέλεσης των εντολών πληρωμής που γίνονται από τους ιδιώτες δικαστικούς επιμελητές. Είναι μια πολύ άδικη μεταχείριση αυτή που επιφυλάσσεται στους βουλγαρούς πολίτες από τις τράπεζες, από τα δικαστήρια, από τις κρατικές αρχές και αυτό είχε τραγικές συνέπειες στις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων. Η Βουλγαρία θα πρέπει να εφαρμόσει ορθά, ορθά την οδηγία 93 κάθετος 213 για, το, για τα δικαιώματα του καταναλωτή επίκυνται νέες προσφυγές. Ο διάλογος με τις βουλγαρικές αρχές είναι εν εξελίξη και γι' αυτό θέλουμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γιάρ, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, να ευχαριστήσω τους αναφέροντες ε, για την πολύ εμπεριστατωμένη παρουσίασή τους ε, εκ των υστέρων. Όταν τα βλέπει κανείς, βλέπει ότι εκεί υπάρχει μοίρα πολλών ανθρώπων που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Άνθρωποι που έχουν αδικηθεί, που χάσαν το σπίτι τους. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ για το πόσο πραγματιστές ήσασταν στην παρουσίαση του προβλήματος. Από την άλλη... Ε, ένα πράγμα που μάθαμε στο σχολείο και μπορεί να έχω και λάθος είναι ότι οι πιστωτέ ε, και οι δανειολήπτες είναι σε μια συμβίωση, έχουν την ίδια μοίρα. Οι τράπεζε ε, στι ε, εποχέ των παχιών αγελάδων είναι πιο γενναιόδορε. Στην πατρίδα μου υπήρξε ένα σοκ στι αρχές του 2000 όταν είδαμε τότε πόσους τίτλους πούλησαν οι τράπεζες χωρίς να το γνωρίζουν καν οι ιδιοκτήτες. Υπήρχαν κάποια ε, οικονομικά προβλήματα, πήγαιναν ε, στην τράπεζα, ε, βάζαν υποθήκη και μετά έχαναν την ιδιοκτησία τους. Στην πατρίδα μου λοιπόν μετά από αυτό βελτιώθηκε ε, μια σειρά νόμων και υπήρξε καλύτερη προστασία των καταναλωτών. Τώρα, συγκεκριμένα για τις αναφορές, ε, πραγματικά είδαμε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών και καλό θα είναι να μείνει ανοιχτή, να μείνουν ανοιχτές οι αναφορές. Το πρόβλημα που βλέπω εδώ και θα ήθελα να βοηθήσω τους συναδέλφους και να με βοηθήσουν, ε, το είπε και η Κομισιόν για την διαδικασία επί παραβάση, όμως, το βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αρκετά γρήγορες οι διαδικασίε. Αυτή είναι μία από... Ε, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε, ότι ε, ζητάμε από την Κομισιόν να κάνει περισσότερα. Ε, πολλές φορές ακόμα και αν το θέλει δεν μπορεί. Ας πούμε στην πατρίδα μου, ας πούμε... Ε, ε, πολλές φορές έπρεπε ε, να πληρώσουν άνθρωποι πρόστιμα ακόμα και 870 ευρώ την ημέρα και έβλεπες ότι ε, δεν μπορούσε κανείς να δράσει γρήγορα ώστε να προστατεύσει τους πολίτες. Ούτε καν τους ίδιους τους πολίτες η κυβέρνηση της Γερμανίας δεν μπορούσε να καλύψει. Πολλές φορές χρειάζεται ένα μορατόριο, να υπάρχει ένα stop για να μπορεί κανείς με ησυχία να συζητήσει ε, τους νέους ε, νόμους. Ε, η Κομισιόν λέει να ένας νέος νόμος, πρέπει να δούμε τι γίνεται εκεί και οι αναφέροντες λένε ότι πρέπει να υπάρχει μια βελτίωση που να γίνει άμεσα. δεν είναι αρκετή η δουλειά που γίνεται. Δεν αρκεί αυτό που λέει λοιπόν η Κομισιόν. Άρα καλό θα είναι να μην είναι ανοιχτή να μείνουν ανοιχτές οι αναφορές, ε, για να υπάρξει ένα μορατόριο, για να μπορούμε να έχουμε χρόνο να σκεφτούμε πώς ακριβώς θα πρέπει να προχωρήσουμε στις απαλωτριώσεις περιουσιών, γιατί πραγματικά ε, το δικό μου coming out είναι ότι ε, οι τράπεζες δεν είναι πάντοτε ε, οι καλύτεροι, ε, ας πούμε, εταίροι των πιστωτών. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Κύρτον έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες και τις αναφέρουσες διότι ήρθαν και υπέβαλαν αυτές τις αναφορές. Το γεγονός ότι είναι μεγάλος αριθμός των αναφορών για το ίδιο ζήτημα δείχνει ότι Υπάρχει συστηματικό πρόβλημα που πρέπει να εξεταστεί και να λυθεί. Και το είπε αυτό και η Επιτροπή. Έχοντας ακούσει λοιπόν όλους τους αναφέροντες, με εκπλήσει η έλλειψη δράσης και από την άλλη χαίρομαι που ακούω από την Επιτροπή τις διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει για τη διαδικασία επί παραβάση και την συνεργασία με τις βουλγαρικές αρχές. Η Επιτροπή μας όμως έχει συμβάλει στο παρελθόν πολύ σε τέτοιου είδους ζητήματα για την προστασία των καταναλωτών, για τα δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια, τα στεγαστικά, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μεταξύ άλλων. Στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία αφιερώσαμε πολύ χρόνο για να λύσουμε το θέμα στην Ισπανία. Είχαμε ψήφισμα στην Ολομέλεια. Εξετάσαμε εκ του στον τρόπο με το οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία για ε, τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια στην ε, Ισπανία. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν υπάρχει δέσμευση για να λυθεί το ζήτημα σε χώριο επίπεδο, Πολύ συχνά όταν χύνεται φως ένα θέμα από πηγές έξω από τη χώρα, επιταχύνεται ο ρυθμός επίλυσης του προβλήματος στο εσωτερικό της χώρας. Συμφωνώ λοιπόν με τους προηγούμενους ομιλητές, πρέπει να παραμείνει οπωσδήποτε ανοιχτή η αναφορά, πρέπει να παραπεμφθεί το θέμα και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και αλλού, ε, γιατί τους ενδιαφέρουν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η προστασία του καταναλωτή και πρέπει και οι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές συναρμόδιες να εξετάσουν το θέμα. Ενδεχομένως αξίζει να υπάρξει αποστολή διερευνητική από την Επιτροπή Αναφορών Επιτόπου στη Βουλγαρία για το θέμα αυτό, για να δούμε ε, όχι μόνο θέματα που άπτονται της αρμοδιότητάς μας για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται όλα αυτά επί από τους ιδιώτες δικαστικούς επιμελητές. Δηλαδή, μια εξέταση από πηγές έξω από τη χώρα μπορούν να επιταχύνουν ε, την επίλυση μιας κατάστασης αρκετά επαχθούς για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ο καθένας πρέπει να νιώθει περισσότερο ασφαλή στο σπίτι του παρά οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι το φυσικό, το φυσιολογικό και το να φοβάται κανείς και να νιώθει ανασφάλεια ότι θα τον πετάξουν έξω από το σπίτι του και θα το βγάλουν είναι ένα συνέστημα φοβερό και θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη στη δική μας ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Παραπέμπω λοιπόν αυτό το αίτημα στους συντονιστές ε, να δούμε ποια συνέχεια πρέπει να δοθεί. Να κάνουμε μια διερευνητική αποστολή, να υποβάλουμε προφορικό ερώτημα στην Ολομέλεια. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοθεί συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Άουκεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους αναφέροντες και τις αναφέρουσες. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να κάθεται κανείς εδώ και να ακούει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ε, τα παρακολουθώ, συμφωνώ και προσθέτω το εξής η Επιτροπή θα πρέπει να τα ακούσει όλα αυτά πολύ προσεκτικά. Δεν αρκεί να γίνουν κάποιες ε, τροπολογίες μικρές. Δεν αρκούν αυτά. Είναι συστηματικό το πρόβλημα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη εξουσία, με μεγαλύτερη ισχύ. Στηρίζω όλα αυτά που προτάθηκαν. Ευχαριστώ τους αναφέροντες και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να δείξει ότι είναι καλή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, ε, για τους πολίτες, τους φυσιολογικούς καθημερινούς πολίτες και σε χώρες που ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ευχαριστώ κύριο Σλοβάκοφ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι έχουμε όλοι καταλάβει πόσο τεράστιο, πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι σαφές. Διαβεβαιώνω τους αναφέροντες επ' αυτού. Όσοι αγωνίζονται για τη δικαιοσύνη και για τα δικαιώματα των πολιτών, αυτό το αντιλαμβάνονται πλήρως. Εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το καθήκον, την υποχρέωση να βρούμε λύση δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση κατά αποκοπήν. Σήμερα να βγάλουμε ένα φυρμάνι και αύριο κάποιο άλλο. Κατά περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει επανειλημμένος. Μπορεί να αποφασίσει να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Ως Βουλγαρός βεβαίως δεν με ικανοποιεί να υπάρχει διαδικασία επί παραβάση. Ε, νομίζω ότι οι συμβάσεις αυτές έχουν ε, αθέμητους είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί και εγώ θα ταχθώ στο πλάι των αναφέροντων και θα πολεμήσω μαζί τους, θα αγωνιστώ για να δοθεί ένα τέλος και να βρεθεί μια λύση σε αυτά τα προβλήματα. Επιμένω προσωπικά και επιμένω και εξ ονόματος της ομάδας του ECR, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή. Ευχαριστώ τους αναφέροντες. Ο κύριος Νικολάη Λαπανό. Αν και ε, δεν συμμεριζόμαστε πλήρως τις απόψεις όλων των ετούντων. Νομίζουμε ότι περιγράφουν ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο επιδρά όχι μόνο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη Βουλγαρία, αλλά επιδρά επίσης σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και στη δική μου χώρα, στην Ελλάδα. Θέλω να επισημάνω στους ε, συναδέλφους στην Επιτροπή Αναφορών ότι εχθές εκκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικών πληστηριασμών στην Ελλάδα, βγάζοντα στο σφυρί 120.000 πρώτε κατοικίε. Κατά την άποψή μα, αυτό δεν είναι, μια, ε, δεν είναι κάτι το οποίο σχετίζεται μόνο με τον νόμο που εφαρμόζει το κάθε κράτο στην κάθε χώρα, καθώ συνδέεται με τη συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίο δημοσιονομικό χώρο για να βρεθεί χρειάζεται να λυθεί ένα πολύ βασικό πρόβλημα, το οποίο είναι αυτό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, των κόκκινων δανείων. Τα μέτρα τα οποία παίρνονται δεν ε, κοιτούν να στραφούν ενάντια στις οφειλές των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, αλλά κοιτούν να στραφούν ενάντια στους εκατοντάδες χιλιάδες μικρόφιλέτες και εφαρμόζουν μέτρα τα οποία είναι η δέσμευση των καταθέσεων, των καταθετικών τους λογαριασμών, των συνταξιοδοτικών λογαριασμών, των ε, λογαριασμών των, των μισθών τους, ο πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Άρα λοιπόν έχει και μεγάλη δόση ε, υποκρισία η τοποθέτηση της Κομισιόν, αφού για παράδειγμα στην ελληνική περίπτωση που συμβαίνει τώρα όπως και στη βουλγάρικη ή και στην ισπανική περίπτωση πριν από χρόνια, ήταν τα μέτρα τα οποία η Κομισιόν σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις εφάρμοσε, τα οποία οδήγησαν στην κατάσταση την οποία είπαν να βγουν στο σφυρί εκατοντάδες χιλιάδες πρώτες κατοικίες. Κατά την άποψή μας πρέπει να μείνει ανοιχτή Πρέπει να μείνουν ανοιχτέ οι αναφορέ που καταθέτουν οι ετώντε. Και κατά την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματο τη Ελλάδα, αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα, σε κάθε χώρα και γενικότερα, είναι πραγματικά να νομοθετηθεί η απαγόρευση του πληστηριασμού τη πρώτη κατοικία, η απαγόρευση τη κατάσχεση και τη δέσμευση των καταθετικών συνταξιοδοτικών και μισθολογικών λογαριασμών από τι τράπεζε και τα ιδιωτικά funds. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η πρόεδρο, Κύριε Κάνεφ, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Είμαι βούλγαρος δικηγόρος και σας επιβεβαιώνω. Πρόκειται για πάγιο πρόβλημα της χώρας μας. Δεν πρόκειται περί μεμονωμένων υποθέσεων πηγή του προβλήματος είναι μια πάρα πολύ ε, άνηση νομοθεσία. Σχετίζεται αυτό και με τη θέσπιση της κατά την προηγούμενη τραπεζική κρίση. Ε, τελικά ε, απέκτησαν πάρα πολύ ισχύ οι χρηματοπιστωτικές ε, ε τράπεζες, οι τράπεζες γενικότερα και ε, οι άλλοι οργανισμοί που δανείζουν τους καταναλωτές εναντί αυτών. Δηλαδή υπάρχει αυτή η άνεση σχέση. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως έχει αρχίσει τη διαδικασία παραβάση κατά της χώρας. Τώρα, όσον αφορά τι προτινόμενε τροποποίησει τη ε, νομοθεσία μα, κατά τη γνώμη μου δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Αλλά θα πρέπει τώρα να λάβουμε υπόψη και κάτι άλλο. Τι γίνεται με την ε, δικονομία, μήπως παραβλάπτει τα συμφέροντα των ε, διαδίκων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για πρέπει να το δούμε καλύτερα. Νομίζω είναι σωστό να γίνει μια ε, διερευνητική αποστολή και επίσης να ασχοληθούν και άλλες συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Και δεν μιλώ για τις ε, επιτροπές που ασχολούνται με οικονομικά θέματα, αλλά αυτές που ασχολούνται με νομικά θέματα, όπως η Νομική Επιτροπή, η Επιτροπή ε, πολιτικών δικαιωμάτων. Θα πρέπει να επιτέλους να υπάρχουν δίκαιες δίκες στη χώρα. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Αντανόκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, λέει η κυρία Ντανόκα. Να μην επαναλάβω αυτά που προείπαν οι συνάδελφοι. Βεβαίω και είναι σωστό να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Πάντως, ε, φάνηκαν πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία τα οποία ακούστηκαν σήμερα σε σχέση με την ε, δίωξη των δικηγόρων που είναι συνήγοροι των ε, αδικουμένων. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει αυτό να το προσέξει ιδιαίτερως. Δεν έχει αναφερθεί αυτό το γεγονός στα έγγραφα που έχουν υποβληθεί. Επίσης, θα πρέπει οι παρόντες δικηγόροι ακριβώς για τη δίωξή τους να υποβάλλουν αναφορά. Ότι δηλαδή δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως συνήγοροι υπέρ των πελατών τους. Βεβαίως και να γίνει μια ερευνητική των πραγμάτων ε, αποστολή. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Τώρα, και ο Ζαμπάσκη έχει το λόγο. Πρόεδρε, λέει ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, ευχαριστώ και τους ε, αναφέροντες αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια σειρά αναφόρων που έχουν υποβληθεί και από όλες προκύπτει κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Κάποιοι φιλέτε, κάποιοι που πήραν κάποιο ενυπόθηκο δάνειο, τώρα έχουν βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Έχουν χάσει ε, τα σπίτια του, ε, τώρα είναι οφειλέτε. Είναι θέμα μόνο πόλη των τραπεζών. Επίση υπάρχουν και κάποιε ε, άλλε εταιρείε στην Βουλγαρία που κάνουν τα ίδια πράγματα όπως και οι τράπεζες, όπως μια εταιρεία που αφορά τη θέρμανση ε, χρησιμοποιούν και ε, αυτοί τους ιδιώτες ε, δικαστικούς κλητήρες και οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Έχουν μια σειρά προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Τα ακούσατε και από τους αναφέροντες, όμως ότι αυτό έπεσε στο κενό έγιναν δραστηριότητες λόμπι και για άλλους λόγους δεν έγινε τίποτα. Ποιοι είναι όμως οι άλλοι λόγοι. Αναφέρθηκε η ερευνητική των πραγμάτων αποστολή, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Βεβαίως θα πρέπει να απευθύνουμε και κάποιες επιστολές στη χώρα. Πάντως αυτή τη στιγμή οι τράπεζε στη Βουλγαρία δεν είναι βουλγαρικές. Όλε αυτέ τι τράπεζες που χρησιμοποιούν τους ιδιώτες ε, δικαστούς κλητήρες είναι γαλλικέ, ταλικές, γερμανικέ, δεν είναι βουλγαρικές. Οι δικηγόροι που έρχονται δεν μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Πρόκειται για αλλοδαπέ τράπεζε. Οπότε, συνάδελφοι, θα πρέπει να απευθυνθούμε και ε, στην ε, ε, μητρική εταιρεία αυτών των τραπεζών να σταματήσουν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Είναι δεσπόζουσα και καταχρηστική η θέση αυτών των τραπεζών, έχουν διαφέρει και τους πολιτικούς ε, που δουλεύουν για αυτές τις τράπεζες. Πάντως σας επενδυμίζω ότι υπάρχουν ε, κάποιοι που έχουν αυτέ τις τράπεζες. Άρα οι επιστολές θα πρέπει να και σε εκείνους. Να γίνει ένα μορατόριο, να παγώσει η διαδικασία αυτή της κατάσχεσης των ε, σπιτιών. Να σταματήσουν να έχουν οι τράπεζες αυτή τη δεσπόζουσα καταχρηστική θέση. Ε, βέβαια θα πρέπει να υπάρξει τροποποίηση τη εθνική νομοθεσία. Και φυσικά οι αναφέροντες ε, αξίζουν τι ε, προστασίε μας. Άρα να μείνουν οι αναφορές ανοιχτέ. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ακούσαμε όλους τους αναφέροντες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τους ε, συναδέλφους της Επιτροπή. Είναι ομόφωνη η γνώμη, οπότε προτείνουμε να μείνουν ανοιχτέ όλες οι αναφορές και να αποστείλουμε κάποια δυναμική επιστολή στη Βουλγαρία και να πούμε ότι προβληματιζόμαστε και ανησυχούμε, θέλουμε να υπάρξει προστασία του καταναλωτή και επίσης θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα παγώματος των κατασχέσεων και εξώσεων. Οπότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να μας αναφέρει σχετικά και να μας πει τι γίνεται και με την διαδικασία επί παραβάση, αλλά και τι γίνεται με την προσπάθεια τροποποίησης της νομοθεσίας από πλευρά του Κοινοβουλίου και του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου. Να υπάρξει μια προστασία των καταναλωτών. Οκτώβριο-Νοέμβριο θα γίνει η έγκριση του νομοσχεδίου. Οπότε πέστε μας τι γίνεται και με την αγωγή κατά της χώρας και τι γίνεται με την ε, νέα βουλγαρική νομοθεσία επίσης. Ήδη έχουμε απευθυνθεί στην ΙΜΚΟ, εμείς ως Επιτροπή Αναφορών. Οπότε θα τις υπενθυμίσουμε τα των αναφορών αυτών, πρόκειται να τις ε, διαβιβάσουμε και στην Οικονομική Επιτροπή. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και 24 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου θα δούμε τι θα γίνει ε, με αυτή την ε, αποστολή που αναφέρθηκε για να γίνει το πρώτο εξάμεινο του 20. Και επομένως θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τι εξελίξει αυτές τις αναφορές από τη Βουλγαρία. Και πάλι ευχαριστούμε τους ε, αναφέροντες που ήρθαν σήμερα εδώ. Από κοντά, από κοντά θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη. Και τώρα προχωρούμε. Η επόμενη αναφορά. Προέρχεται από πρόσωπο γκρικής ηθαγενείας. Ε, έχουν υπογράψει και άλλοι 10.000 σχετικά με καταχρηστικού συμβαστικού όρου δανείων σε ξένο νόμισμα στην Ουγγαρία. Δεν παρίσταται ο αναφέρον. Τι είπατε? Α, όχι, όχι συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, είναι εδώ ο αναφέραν. Πολύ ωραία. Έχετε πέντε λεπτά για να μας μιλήσετε. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους ε, των ε, συμπολιτών μου δεν είμαστε εδώ για να έχουμε κάποια ειδική μεταχείριση, αλλά για να κερδίσουμε την ίση μεταχείρισή μας. Κυρίες και κύριοι, φανταστείτε να πηγαίνετε στην τράπεζα για ένα δάνειο και παίρνετε δάνειο στο δικό σας εθνικό νόμισμα, αλλά τελικά το δάνειο καταγράφεται σε ξένο νόμισμα, παρόλο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας. Αυτό είναι δυνατό μόνο αν γίνει μετατροπή ε, στο ξένο νόμισμα τη στιγμή που γίνεται η λήψη του δανείου. Έτσι μπορεί η τράπεζα ε, δεν μπορεί η τράπεζα ε, να αυθαίρετα να αυξάνει το επιτόκιο και να παίρνει προμήθειες από τις ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες. Μετά από πολλά χρόνια λοιπόν πηγαίνει στο δικαστήριο και λες ότι είχες άδικη μεταχείριση και στο δικαστήριο μαθαίνεις ότι δεν ήσουν καν αντισυμβαλόμενος σε αυτή τη συναλλαγή. Ε, Πιλάμε για χρήματα ε, πολλά ευρώ σε μηνιαίες δόσεις και το δικαστήριο σου λέει ότι το Εθνικό Κοινοβούλιο θα πάρει ε, αποφάσεις ε, για τα αυτά τα χρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, τα οποία θα θεωρηθούν ότι είναι υπερβάλλουσες ε, καταβολές. Όμως, ήδη έχεις καταδικαστεί ότι δεν έχεις πληρώσει. Οι παραπάνω αυτές, τα παραπάνω αυτά χρήματα που έχεις δώσει σου επιτρέπουν με να, να καλύψεις κάποια ποσά, όμως δεν μπορείς να πάρεις τα χρήματα πίσω. Επίσης καταγγέλλεται η σύμβαση και ξεκινάνε οι διαδικασίες ε, εκτέλεσης. Ε, επίσης το Κοινοβούλιο βγάζει και άλλο νόμο που λέει ότι θα ε, μετατραπεί και θα παγώσει στο ουγγρικό νόμισμα το δάνειό σου και το κεφάλαιο και η τοκη μετα μετά από 5-10 χρόνια αποπληρωμής του δανείου θα είναι τρεις φορές παραπάνω από ό,τι αρχικά είχε λάβει ως δάνειο. Στη συνέχεια, το ανώτατο δικαστήριο αποφασίζει ότι αυτό που πήρες ήταν μια υποχρέωση χρέους παρόλο που εσύ δεν έδωσες δάνειο στην τράπεζα, να πάρεις δάνειο θελες Είναι άλλο πράγμα από ότι είναι η αποπληρωμή δανείου αυτό στην νομοθεσία. Τι θέλανε λοιπόν να κάνουν, να καλύψουν το γεγονός ότι αδίκως χρεώθηκε σε τις εμπορικές αυτές προμήθειες της τράπεζας για τις συναλλαγές. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν στην Ουγγαρία είναι η ληστεία του αιώνα. Έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια στο ουγγρικό δικαστικό σύστημα και ε, γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ και σας ζητούμε να εφαρμόσετε την ε, οδηγία 93-13 και ζητούμε άμεση εφαρμογή, να ε, σταματήσουν ε, οι ε, παλαιτριώσεις και να αποζημιωθούν αυτοί που έχασαν την ιδιοκτησία τους. Θα θέλαμε να βοηθήσετε τους Ούγκρους πολίτες να ξανακερδίσουν την αξιοπιστία τους ενώπιον του ευρωπαϊκού νομικού συστήματος. Εγώ προσωπικά είχα 47% παραπάνω ποσά να πληρώσω στις μηνιαίες δόσεις μου. Το αναγνωρίζει και η τράπεζα. Έχει παρόλα αυτά ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης εναντίον μου. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες, υπάρχουν χιλιάδες μάλλον άνθρωποι οι οποίοι ε, έχασαν τις περιουσίες τους, ε, είναι σε κίνδυνο και πολλοί έχουν φύγει και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να μπορέσετε να μας βοηθήσετε. Παρακαλώ αφήστε ανοιχτή την αναφορά και κάντε ό,τι μπορείτε προκειμένου αυτές οι παράνομες εξώσεις ε, και διαδικασίες εκτέλεσης να σταματήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Τη σειρά έχει η Επιτροπή, ο κύριος Πίτερ Μπίσοπ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο ε, αναφέρον αναφέρεται σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν δάνεια σε ξένο νόμισμα. Ενυπόθηκα δάνεια ε, σε ξένο νόμισμα με υψηλό ε, κίνδυνο, υψηλή επικίνδυνοτητα σε σχέση με την ε, εξέλιξη της συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η οικονομική κρίση, η χρηματοπιστωτική κρίση από το 2008 και μετά οδήγησε ε, σε υποτίμηση νομισμάτων στις, Ανατολικ... στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Έπρεπε ε, να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά ε, από ό,τι θα πλήρωναν αν τα δάνεια ήταν στο τοπικό τους ε, νόμισμα. Και αυτό ακριβώς έγινε και στην περίπτωση του αναφέροντος που έχει αύξηση κατά 50% στις δόσεις. 2014 κάθετος 17 είναι η οδηγία που αφορά στις πιστώσεις και λέει ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μειώνουν το συναλλαγματικό κίνδυνο είτε δίνοντας στους καταναλωτές το δικαίωμα να μετατρέπουν σε άλλο νόμισμα ή μέσα από άλλες διευθυντήσεις π.χ. ανώτατα όρια. Αυτή η οδηγία για τα τυπώθηκα δάνεια όμως δυστυχώς εφαρμόζεται μόνο ε, σε δάνεια που δόθηκαν μετά την 21η Μαρτίου του 2018, όχι σε αυτά που δόθηκαν πριν την οικονομική κρίση μετά, στην επαύριό Έτσι λοιπόν, ε, όσοι πήραν δάνειο πριν από το Μάρτιο του 2016 εμπίπτουν στο Γενικό Καταναλωτικό δίκαιο, ας πούμε, την οδηγία για τις ε, καταχρηστικές ε, διατάξεις και όρους δανείων και τις ε, καταχρηστικές, άδικες ε, πρακτικές, εμπορικές πρακτικές που ήταν ας πούμε τρόπος πώλησης αυτών των δανείων από τις τράπεζες. Η οδηγία για τους άδικους όρους καταναλωτικών συμβάσεων είναι ακριβώς αυτό που αφορά τον αναφέροντα. Τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη εκδώσει αποφάσεις για την ερμηνεία και την εφαρμογή αυτής της οδηγίας ε, όσον αφορά σε δάνεια σε ξενονόμισμα. Πολλά από τα αιτήματα προέκυψαν από ουγγρικά δικαστήρια. Τα, αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου συνεισέφεραν ιδιαίτερα στην διαλεύκανση της νομικής κατάστασης, ειδικά η απόφαση 4η Μαρτίου του 2019, μια πρόσφατη υπόθεση, είναι πολύ σημαντική. Τονίζει ότι η βασική αρχή της οδηγίας ε, είναι ένας όρος ε, ο οποίος ε, θεωρείται άδικος από δικαστήριο, δεν δεσμεύει τον καταναλωτή. Το Εθνικό Δικαστήριο Αυτεπαγγέλτος θα πρέπει να καταργεί αυτούς τους όρους, να ακυρώνει τους όρους αυτούς και να συνεχίζει η υπόλοιπη σύμβαση όσο έχει. Αν δεν μπορεί μια σύμβαση να συνεχίσει χωρίς αυτόν τον όρο, θα πρέπει συνολικά η σύμβαση να θεωρείται άκυρη. Αυτό είναι ένα θέμα που μόνο ένα εθνικό δικαστήριο μπορεί ε, για κάθε υπόθεση να κρίνει. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Στη δική του υπόθεση ε, για το θέμα αυτό μίλησε για την νομοθεσία που η Ουγγαρία υιοθέτησε το 2014 για αυτά τα δάνεια σε ξένο νόμισμα. Σύμφωνα με αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μία από τις διατάξεις της Ουγγρικής νομοθεσίας ε, ε, εναντιώνεται στις διατάξεις της οδηγίας για τις άδικες διατάξεις συμβάσεων, διότι δεν επιτρέπουν στους καταναλωτές να μην δεσμεύονται από τους άδικους όρους ε, ή να δεν επιτρέπει να ακυρώνεται μία σύμβαση όταν ε, δεν μπορεί να ε, συνεχίσει χωρίς τον όρο που είναι άδικος και πρέπει να ακυρωθεί. Αυτές οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήρου και γενικά ο διαρθρωτικός διάλογος με τις Ουγγρικές αρχές μας βοήθησαν να ζητήσουμε πληροφορίες από τις Ουγγρικές αρχές για να δούμε πώς θα εναρμονίσουν την νομοθεσία τους με την Ευρωπαϊκή. Η απάντηση αναμένεται στα τέλη του Οκτωβρίου. 22 Ιουλίου του 2019 εστάλει μία καθοδηγητική ε, ειδοποίηση ε, όπου η Κομισιόν ε, μιλάει σε συγκεκριμένη παράγραφο για αυτά τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και αναφέρεται στη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Παρακαλώ διαβάστε αυτό το έγγραφο, το Guidance Note και θα δείτε ακριβώς, βέβαια αυτό ε, αφορά κυρίως ε, τους εξειδικευμένους επαγγελματίες, ε, δικαστές, δικηγόρους που πρέπει να εφαρμόσουν σωστά τους κανόνες σύμφωνα με την ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τη σειρά έχουν τα μέλη της Επιτροπής μας. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Η ε, κυρία Κύρτον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και πάλι, όπως και στην περίπτωση της προηγούμενης αναφοράς, η ομάδα αναφορών, θα ήθελα να πω τα εξής. Ε, με τους αναφέροντες από τη Βουλγαρία είχαμε μεγάλο αριθμό αναφερόντων στην Επιτροπή, ενώ εδώ έχουμε έναν αναφέροντα που εκπροσωπεί πάρα πολλούς ανθρώπους στην Ουγγαρία. Η διαφορά είναι μόνο αυτή. Η ουσία όμως παραμένει η ίδια. Οι άνθρωποι υπόκεινται σε αθέμητους συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις. Η Επιτροπή μας είπε ότι υπάρχουν σαφείς τομείς όπου δεν τηρείται το ευρωπαϊκό δίκαιο και είναι δική μας ευθύνη και αρμοδιότητα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα αναδείξουμε όλα αυτά, ε, να αναδείξουμε αυτές τις υποθέσεις προστασίας του καταναλωτή και να ε, στείλουμε αυτό το μήνυμα ότι πρέπει και μπορεί ο Ευρωπαίος πολίτης να βασίζεται και να στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την προστασία του, για τα καταναλωτικά του δικαιώματα, ε, για όλα αυτά τα θέματα. σε σχέση με τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια ή με οτιδήποτε άλλο, με οποιαδήποτε άλλη σχέση του με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Περιμένουμε απάντηση των Ουγγρικών Αρχών τον Οκτώβριο, μας είπε η Επιτροπή, ε, όμως ξέρετε πάνω κάτω ποια συνέχεια θα δοθεί. Έχετε κάποιες σκέψεις για το αν θα γίνει η διαδικασία επί και ποια θα είναι τα επόμενα στάδια εάν δεν αποκαταστήσουν ε, το δίκαιο οι Ούκρικες αρχές. Δηλαδή με ενδιαφέρει να μάθω ποια είναι η προοπτική, πώς το βλέπετε, τι θα πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τον Οκτώβριο. Δεν μπορεί να μην ξέρετε ή να μην έχετε κάποια ιδέα. Η σύσταση της δικής μας Επιτροπής είναι να προχωρήσει το θέμα. Όμως, αν η Επιτροπή δεν το ολοκληρώσει, τότε ε, να παραμείνει αναφορά να σταλεί και στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και ΙΜΚΟ για τα, τους καταναλωτές, για τα οικονομικά, γιατί είναι συναρμόδιες και τις αφορά. Με ενδιαφέρει λοιπόν να μάθουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς βλέπει να εξελίσσεται το χρονοδιάγραμμα και πώς ε, στοχεύει να κινηθεί μετά τον Οκτώβριο και την απάντηση των Ουγγρικών αρχών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δουράκη μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Ντούδα και μετά η Επιτροπή. Θα αντικαταστήσω τη συνάδελφο Σιμακοπούλου και θα παρουσιάσω ε, τη σύντομη γνωμοδότησή της. Και διαβάζω. Παραθέτω τα εξής. Οι αθέμητες συνθήκες και περιστάσεις ε, για τα διάφορες συμβάσεις τις καταναλωτικές, ε, ε δανειακές συμβάσεις με καταχρηστικούς συμβατικούς όρους, Όλα αυτά ρυθμίζονται από την οδηγία, από την οδηγία 2.14 κάθετος 17 και αυτά είναι τα καλά νέα. Ε, έχουν, αφορά παρόλο που τα δάνεια που έχουν συναυθεί πριν το Μάρτιο του 2016 δεν διέπονται από αυτή την οδηγία, αλλά από την οδηγία 93 κάθετος 13 για τις αθέμητες ε, συνθήκες και όρους και περιστάσεις στο δίκαιο του καταναλωτή και σε τέτοιου είδου συμβατικέ υποχρεώσει. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται και μεριμνά για τη σωστή εφαρμογή των δύο οδηγιών στην Ουγγαρία και αυτό θα βελτιώσει την, την κατάσταση των δανειοληπτών. Και γι' αυτό θέλουμε να κλείσει η αναφορά. Δεν έχουμε άλλο μέλος τη επιτροπή μας που θέλει να πάρει το λόγο και γι' αυτό δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Thank you, Madam Chair, and also thank you for um, the clarification question from uh, um, the Honourable Member. Σας ευχαριστώ. Ε, θα προσπαθήσω να απαντήσω στα διευκρινιστικά ερωτήματα. Στην απόφαση ε, του Μαρτίου, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ανέφερε ξεκάθαρα Πού έγκυται το συγκεκριμένο πρόβλημα στην Ουγγρική νομοθεσία. Εντόπισαν μια συγκεκριμένη διάταξη σε έναν από τους εφαρμοστικούς νόμους της Οδηγίας 2014 και έδωσαν σαφείς γραμμές κατευθυντήριες στον Ούγκρο νομοθέτη για το πώς μπορεί να αποκατασταθεί το δίκαιο και να λυθεί το πρόβλημα. Το δικαστήριο θεώρησε ότι συνολικά η Ουγγρική νομοθεσία, γιατί είναι τρεις οι νόμοι που ε, ε, είναι συναρμόδιοι, φαίνεται να είναι τρόποντινά συμβατεύστο, συμβατό. Το σύνολο λοιπόν της Ουγγρικής νομοθεσίας φαίνεται να είναι την συμβατό με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο για αυτά τα ζητήματα. Εκτός από αυτό το σημείο που χρήζει επιδιόρθωση ή αποκατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να σας πούμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε στη συνέχεια. Πρέπει να δούμε πρώτα τι θα απαντήσουν οι Ουγγρικές αρχές τον Οκτώβριο. Εάν προτίθεται να ε, παράγουν νομοθετικό έργο, αν έχουν ήδη υιοθετήσει νομοθετική πρωτοβουλία για να αφαιρεθεί αυτό το εδάφιο στην Ουγγρική νομοθεσία που δημιουργεί και το πρόβλημα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα περιμένουμε να εγκριθεί αυτή η νομοθεσία ε, αν προτίθενται να την φέρουν προς ψήφιση. Από εκεί και πέρα, από τεχνικής πλευράς, ίσως προτείνουμε στην Επιτροπή να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάση. Όμως το να ξεκινήσει μια διαδικασία επί είναι απόφαση του σώματος των, επιτρόπων. Και η συνέχεια που θα δίδεται σε διαδικασία επί κάθε φορά είναι απόφαση του σώματος των επιτρόπων. Άρα πρόκειται για πολιτική απόφαση και δεν μπορώ να την προβλέψω και να την υποδικάσω. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε το θέμα στενά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Ο αναφέρον έχει το λόγο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή αυτά που είπε ο κύριος και με το μεγάλο του ενδιαφέρον. Νομίζω ότι ζούμε σε παράλληλους κόσμους. Η αναφορά δεν έχει να κάνει με την αλλαγή ε, του νομίσματος. Ε, ήδη το δικαστήριο είπε ότι είναι αθέμητη η όρη, είναι καταχρηστική συμβατική όρη. Ψηφίστηκε η νέα νομοθεσία, αλλά δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. 1.900.000 δανειακές συμβάσεις είναι αυτές. Οι τράπεζες έστειλαν ένα έγγραφο στους πολίτες ε, που έλεγε πόσα χρήματα ήδη όφυλαν, πόσα χρήματα είχαν ήδη καταβάλει και μέρος αυτών είχε, ε, το είχαν πάρει καταχρηστικά. Πάρα πολλές από αυτές τις συμβάσεις έχουν ήδη λήξει και λυθεί και προωθήθηκαν για άμεση εντολή πληρωμής ή αλλιώς ε, εκένωση και εξώδικο για να βγάλουν τον κόσμο από τα σπίτια του. Κι εγώ πήρα ένα τέτοιο χαρτί ότι δηλαδή μου παίρνουν την ιδιοκτησία μου. Δεν μπόρεσα να πληρώσω φόρους ούτε στην Ουγγαρία ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 7 χρόνια. Δεν μου επιτρέπουν να αποκτήσω αυτοκίνητο στο όνομά μου. Έχω ένα χαρτί όμως που μου έχουν ληστέψει και ε, ουσιαστικά μου λένε 12.000 ε, ε, ελβετικά φράγκα. Δεν υπάρχει Τίποτα που μπορώ να κάνω. Μιλούμε για το μέλλον χιλιάδων οικογενειών. Δεν είναι το θέμα ότι δεν δόθηκαν σαφή στοιχεία οι πληροφορίες ή δεν ενημερώθηκαν σωστά οι καταναλωτε Το δικαστήριο ήταν πολύ συγκεκριμένο. Οι, οι όροι ήταν αθέμητοι. Αυτό το αποφάσισε το δικαστήριο. Και παρόλα αυτά αγρόνα αγοράζουν και συνεχίζουν να βγάζουν τον κόσμο από τα σπίτια του. Ευχαριστώ. Η προεδρο ευχαριστώ το αναφέροντα, διότι ήρθε εδώ σήμερα, άκουσα το αναφέροντα τα μέλη της Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επομένως ως Προεδρείο ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και να σταλεί εστάλει το Μάρτιο του 19 στην Επιτροπή ΕΚΟΝ και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και θα την ξαναστείλουμε. Ζητούμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για την απάντηση των κρατικών αρχών ή της κυβέρνησης της Ουγγαρίας τον επόμενο Οκτώβριο, για να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα εκ του και να δούμε ποια συνέχεια θα δοθεί. Εκτός μικροφώνου η Πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν και κλείνουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Πάμε στο σημείο 21. Αναφορά υπεριθμών 0692 κάθετος 2018 της Καταλίνα Θέρδα Πόνς, Ισπανικής Εθαγένειας, για την εφαρμογή του κανονισμού 261-2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς, σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματέωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης. Και έχουμε και την αναφορά 0727 του 2018 ενός πολίτη γερμανικής ηθαγένεια για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωση για άρνηση επιβίβαση, ακύρωση πτήσεων ή μεγάλες καθυστερήσεις. Κανένα από τους δύο αναφέροντες δεν είναι παρόν και γι' αυτό δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Όσον αφορά αυτές τις αναφορές, αφορούν αυτόν τον κανονισμό για τα ε, δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Πρώτα απ' έχουμε 692 του 18. Αυτή η αναφορά αφορά αυτή την ε, πρακτική του overbooking που κάνουν οι αεροπορικές ε, εταιρείες και για μια σειρά πτήσεων ε, του 18 λέει η αναφέρουσα ότι πέστη στην Ισπανία ε, αυτή την πρακτική του overbooking. Δεν έχω άλλες λεπτομέρειες, οπότε πρόκειται για μια πρακτική που δεν είναι παράνομη καθε αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις που διέμουν τα δικαιώματα των επιβατών. Ε, ο κανονισμός 261 λέει ότι μια αεροπορική εταιρεία όταν αρνηθεί ε, σε κάποιον την επιβίβαση θα ζητήσει ε, από αυτούς που δεν επιβεβαίνουν να εμπολίσουν το δικαίωμά τους. Τώρα, εάν δεν έχουμε αρκετούς εθελοντές που παρετούνται από τη θέση τους και έτσι να μπορούν να χωρέσει του υπόλοιπου του αεροπλάνο, τότε η αεροπορική εταιρεία μπορεί να αρνηθεί σε αυτού που δεν έχουν προσφέρει, σε κάποιου και να του δώσει ε, αποζημίωση. Και έτσι αυτοί που διάσουν τα χρήματα για εναλλακτικέ λύσει. Ε, θα πρέπει αυτοί οι να εφαρμόζονται. Ε, έχει κρυθεί και έχουμε το άρθρο 14 του κανονισμού θα πρέπει να γίνει επομένω στην εφαρμογή του και θα πρέπει να ε, ενημερώνονται οι επιβάτε σε τέτοια περίπτωση και στο τσεκίνο ότι δεν τους αφήνουν να επιβούν, αλλά ε, και στο γκισέ, e, αλλά και ιντερνετικά όταν πάνε κάνουν το check-in. να αφορά την αποζημίωση. Έχουμε να πούμε ότι στην πρότασή μας του 2001 σε σχέση με τους κοινούς κανόνες για αρρωγή και αποζημίωση σε αυτούς οι που έχουν υποστεί την άνεση επιβίβασης, έχουμε προτείνει υψηλότερη αποζημίωση. Τότε είχαμε πει τα 750 ευρώ για πτήσεις ε, κάτω των 3.500 χιλιόμετρων και είχαμε πει 1.500 ε, ευρώ για πτήσεις πάνω από 3.500 χιλιόμετρα. Ε, αυτό έχει σημασία γιατί η αναφέρουσα λέει ότι η αποζημίωση τώρα είναι 250 ευρώ που το θεωρεί ανεπαρκές ποσό. Αυτό είναι για μέχρι τα 1500 χιλιόμετρα. Οπότε, έτσι, αποζημιούται ο επιβάτης για την ταλαιπωρία και για την απολύχρονη. Πάντως ξεκαθαρίζεται ότι αυτό είναι ένα μήνυμο, ένα ελάχιστο ποσό, το ελάχιστο ε, για τα δικαιώματα των επιβατών που τους αρνούνται την επιβίβαση παρά τη θέλησή τους. Τίποτα στον κανονισμό δεν απαγορεύει στον επιβάτη να επιδιώξει μεγαλύτερη αποζημίωση πέραν των ορίων του κανονισμού Φερρυπίν για τη ζημία που υπέστη ακριβώς επειδή του ειρνήθησαν την επιβίβαση σύμφωνα με το Διεθνές Αστικό Δίκαιο το overbooking είναι όμως ε, κάτι το οποίο δικαιούν το κάνει η εταιρεία, επομένως κάθε αυτό το overbooking δεν ωραία Σήμερα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, περίπου 0,1% των επιβατών υφίστανται την άρνηση επιβίβασης, αλλά ε, σε αυτά τα στοιχεία καλύπτονται και εκείνοι οι επιβάτες οι οποίοι εθελοντικά παρετούνται ε, τις θέσεις τους γιατί προτιμούν να πάρουν αλλιώς τον προορισμό τους ή να πάρουν την αποζημίωση. Το 2013 γίναμε μια πρόταση για τροποποίηση του 261 του 4. Σκοπός ήταν να εξασφαλιστεί η προστασία των δημοτών επιβατών, να ληφθούν υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες των εταιριών. Δεν άλλαξαν τα ποσά της αποζημίωσης. Ακόμα εκκρεμεί η πρότασή μας στο Συμβούλιο και στο Γενοβούλιο γιατί το 2015 μπλοκαρίστηκε η εν λόγω πρότασή μας στο Συμβούλιο. Η πρόεδρο ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα ήρθε η ώρα να λάβουν οι συναδελφοί των λόγων και με ρίξετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Ο κανονισμός του 2001 για το ποσό αυτό είναι ξεπερασμένο μέτρο. Θα πρέπει σήμερα να λάβουμε υπόψη το ότι θα πρέπει η αποζημίωση να ευθυγραμμιστεί με την παρούσα συγκυρία την οικονομική συγκυρία, την ε, νομοθεσία, γιατί πέρασαν αρκετά χρόνια από την θέσπιση σε ισχύ αυτού του κανονισμού. Επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω, ούτως ώστε να προστατεύσουμε περισσότερο τους επιβάτες αυτούς. Έχουν προηγηθεί μία σειρά υποθέσεων σε σχέση με τους δικαιούχους τέτοιων αποζημιώσεων. Επομένως πρόκειται το παλαιού κανονισμού. Άρα θα πρέπει να αναθεωρήσουμε αυτό το νομοθέτημα και να προσαρμόσουμε την αποζημίωση. Ευχαριστούμε πολύ. Λέει στον κύριο Αμερίξ η πρόεδρος. Όλοι τοποθετήθηκαν επομένω και σας προτείνω να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. 2018 έκανε μια έρευνα η Επίτροπη, το 2019 δημοσιοποιήθηκαν αυτά τα ε, προβλήματα, οπότε θα δούμε αυτή η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι έβγαλε, θα τα μελετήσουμε. Ενημερώνθηκαν η ΙΜΚΟ και η ΤΡΑΝ στο Κοινοβούλιο. Επίσης θα ενημερώσουμε και την Νομική Επιτροπή. Γιατί ήδη μελετά μια οδηγία όσον αφορά την νομική εκπροσώπηση. Πάμε τώρα στο σημείο 22. Είναι η αναφορά 165 του 18 του Μάριο Μπέργκερ γερμανικής εθαγενείας και αφορά τον αποκλεισμό των επιβατών σε πτήσεις επιστροφής αν δεν έχουν πάρει την εξερχόμενη πτήση. Δεν έχουμε εδώ τον αναφέροντα, οπότε θα δώσουμε ευθύς αμέσως το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <coughs> Γκίντερ, έτελεχτε ξανά το λόγο. Στην αναφορά 165 του 2018 υπάρχει η, η προσφυγή του αναφέροντος που λέει ότι πήρε ένα εισιτήριο που δεν άλλαζε και έπρεπε να πάρει και την εξερχόμενη πτήση για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την εισερχόμενη πτήση. Επειδή δεν εμφανίστηκε, θεωρήθηκε ότι δεν έχει δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει. Σύμφωνα, <clears throat> λοιπόν, με τον κανονισμό 261, η μη εμφάνιση ε, δεν ε, θεωρείται ότι δεν επιτρέπεται. Έτσι λοιπόν, όταν έχεις μία κράτηση ε, εξερχόμενης και εισερχόμενης ε, πτήσης ε, και δεν εμφανίζεσαι στην εξερχόμενη πτήση, όταν σου αρνηθούν την επιβίβαση στην εισερχόμενη ε, δεν θεωρείται ε, άρνηση επιβίβαση κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού 261. Είναι σημαντικό ο καταναλωτή όμω να ενημερώνεται σαφώ για του όρου μεταφορά τη αεροπορική εταιρεία. Ε, η πραγματικά Επιτροπή έχει επίγνωση των ανησυχιών των καταναλωτών ότι ορισμένοι αερομεταφορείς μπορεί να διευκρινίζουν αόριστα τους όρους μεταφοράς και αν ένας επιβάτης δεν επιβιβαστεί σε κάποια συγκεκριμένη πτήση ενδέχεται να ακυρωθούν η επιστροφή. Επίσης, ε, η Επιτροπή ε, λέει ότι ε, είναι σημαντικό να ενημερώνουν οι πελάτες όταν δεν έχουν σκοπό να εμφανιστούν. Η Επιτροπή έχει επιδιώξει να αντιμετωπίσει το ζήτημα στην πρότασή της για την τροποποίηση του κανονισμού η πρόταση επιβεβαιώνει ότι οι αεροπορικέ δεν μπορούν να αρνούνται την επιβίβαση του ταξίδι επιστροφή του ίδιου εισιτηρίου λόγω του γεγονότο ότι οι επιβάτε δεν είχαν ταξιδέψει στην εξερχόμενη πτήση. Η πρόταση τη Επιτροπή, ε, ε, ε, λοιπόν, ε, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης υπάρχουν και άλλες ε, ρήτρε που θεωρούνται ε, άδικες. Ας πούμε κάποιες αεροπορικές μπορούν, επιτρέπουν τους, τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν ένα κομμάτι της διαδρομής όταν έχουν ενημερώσει εκ των προτέρων. Ευχαριστώ κυρία Αμερίξ. Ξεκινάει ο γύρος των μελών, των βουλευτών μας. Ο κύριος Αμερίξ ε, μάλλον. Ε, κατά τη γνώμη μου, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, διεθνείς δραστηριότητες αυτών των ε, εταιριών θα πρέπει να εξετάσουμε ξανά τους όρους ε, του σχετικού κανονισμού. Έχει περάσει πολύ καιρό από τότε που τον εγκρίναμε. Καλό είναι λοιπόν να αναθεωρήσουμε τις αρχές του ε, προς όφελος των καταναλωτών. Ακούσαμε σήμερα πληροφορίες ε, που δείχνουν πως ε, σε κάποια κράτη-μέλη γίνονται, ε, πραγματοποιούνται αυτές οι πρακτικές, οπότε αυτό καλό θα είναι να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα να ξαναδούμε τον κανονισμό. Εδώ και αρκετό καιρό, λοιπόν, εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός, οπότε καλό θα είναι να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και να φτάσουμε σε συγκεκριμένο συμπέρασμα. Μέχρι να φτάσουμε σε συγκεκριμένο συμπέρασμα. Πολύ ωραία. Αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, έχοντας διαβάσει την αναφορά, έχοντας ακούσει τον αναφέροντα, έχοντας ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόταση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής μας είναι να παραμένει η αναφορά ανοιχτή την στείλαμε στο παρελθόν στην αρμόδια επιτροπή για τις μεταφορές και θα στείλουμε σημείωμα υπενθύμηση στην Επιτροπή Τραν να ασχοληθεί με το θέμα. Ζητούμε από την Επιτροπή επικαιροποιημένες πληροφορίες σε σχέση με την κατάσταση της νομοθεσίας δεν έχουν εγκρίνει την πρόταση Επιτροπής για την τροποποίηση του σχετικού κανονισμού του 2004 και ζητούμε από την Επιτροπή να μας ενημερώσει για όλα αυτά αλλά και για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνούμε λοιπόν στο σημείο 23 της ημερησίας διάταξης αναφορά 0202 κάθετος 2018 από τον Αλφόνσο Ροντρίκεθ Σάντσεθ Ισπανικής Ιθαγένειας για τις ε, πολιτικές διάθεσης θέσεων αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους, οι οποίες χωρίζουν ομάδες και οικογένειες που δεν προσθε... πληρώνουν πρόσθετη χρέωση για κράτηση θέσης. Είναι εδώ αναφέρον ο κύριος Αλφόνσο Ροντρίγκεθ Σάντσεθ και έχει πέντε λεπτά για να μας τα εκθέσει όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μας δίνετε να εμφανιστούμε ε, ενώπιόν σας εδώ στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να σας παρουσιάσουμε τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούν οι αεροπορικέ εταιρείε χαμηλού κόστους και κυρίως η Ryanair και σας ζητούμε να κάνετε τα δέοντα για την υπεράσπιση των ε, πολιτών. Εδώ και κάποια χρόνια έχουν ξεκινήσει έναν το πόλεμο για να προσποριστούν μεγάλο μέρος της αγοράς και μειώνουν την τιμή των πτήσεων, αλλά δεν μειώνουν το περιθώριο κέρδους τους, ενώ μειώνουν τα εισιτήρια. Και ε, ουσιαστικά συνεχίζουν να χρεώνουν για υπηρεσίες οι οποίες ε, ε, σιωπηλά είχαν γίνει αποδεκτές ως μέρος της τιμής του εισιτηρίου. Επομένως δεν βασίζονται ως εμπορική δραστηριότητα στην πώληση των εισιτηρίων αλλά στις παράπλευρες απώλειες για κάποιους που συνεπάγεται η αγορά αυτών των εισιτηρίων οι οποίες μεταφράζονται σε κέρδη για τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Δηλαδή είναι υπηρεσίες χρέωση, οι οποίες ε, ε, δεν... Ε, δεν μιλώ για τις υπηρεσίες χρέωσης οι οποίες μπορεί κανείς να τις αγοράσει ή όχι, να αγοράσει ένα άρωμα στο αεροδρόμιο στο αεροπλάνο. Μιλούμε για διάφορα πράγματα τα οποία ε, είναι πολύ σημαντικά και αν κανείς δεν, ε, δεν προσέξει τη στιγμή που το αγοράζει στο ίντερνετ μπορεί όταν εμφανιστεί στη πτήση του να πρέπει να πληρώσει πάρα πολλά πράγματα επιπρόσθετα, ε, να βρεθεί να μην ξέρει που θα πάει, να μην μπορεί κανείς να πάρει τη βαλίτσα του και το καθεξής. Το ε, των καταγγελιών έχουν να κάνουν με αυτές τις ε, εταιρείε. Δημιουργούν διάφορα προβλήματα στους χρήστες. Δεν μπορώ να τα επαριθμίσω. Είναι πάρα πολλά. Με τη δράση τους το μόνο που κάνουν είναι να πικραίνουν τους χρήστες, να τους χαλάνε το ταξίδι είτε στην αρχή είτε στο τέλος ε, του ταξιδιού τους. Καταρχάς 60 ευρώ ήταν το πρόστιμο αν δεν είχαμε εκτυπώσει μόνοι μας τις κάρτες επιβίβασης. Μετά με τις βαλίτσες, μετά με τις χειραποσκευές, μετά με τα σακίδια και τις, άκες, τη γυναι... τσάντες της Και τώρα, ε, τώρα χωρίζουν και τους ανθρώπους που έχουν κάνει ομαδική κράτηση. Δηλαδή η Ryanair δίνει ξεχωριστές θέσεις αυτόματα, υποχρεωτικά, σε όλους όσους έχουν κάνει ομαδική κράτηση, ανεξαρτήτως του αν είναι φίλοι, γνωστοί ή μέλη της ίδιας οικογένειας, υποχρεωτικά τους χωρίζει και τους ω ως άτομα πλέον για να μην κάτσουν ποτέ μαζί. Και αυτό φαίνεται σε αυτό το μήνυμα και λέει, ότι, και στο μήνυμα ότι αν δεν σε αρέσουν οι θέσει σου μπορείς να τις αλλάξεις. Αυτό το λένε στο ίντερνετ. Όταν όμως φτάνεις καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πληρώσεις από 9 ως 30 ευρώ αναλόγως με τη θέση που διαλέγεις. Δηλαδή ε, χωρίζει οικογένειες με ανήλικα παιδιά ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών την ώρα που εκδίδει τα εισιτήρια. Φανταστείτε να ταξιδεύετε με τον άντρα σας, με τη γυναίκα σας, με τα παιδιά σας και να φτάνετε στο αεροδρόμιο και να έχετε διαφορετικά καθόλου καθίσματα. Ένας ανήλικος, ένα μικρό παιδάκι έχει φοβερό άγχο. Ε, σε περίπτωση επίγοντος κατάσταση κατάστασης στο αεροπλάνο. Να είναι ο ενήλικο στη σειρά 4 ας πούμε και το παιδί στη σειρά 27. Ε, σκεφτείτε μια ε, μητέρα που πάει διακοπέ με το γιο τη 10 ετών και η μία κάθεται μπροστά και ο άλλο η τελευταία σειρά πίσω. Βιώνουν άγχος οι οικογένειε. Οι οικογένειε οι οποίε ταξιδεύουν με άτομα με αναπηρίε ή με άτομα με ψυχολογικά προβλήματα ε, και να είναι υποχρεωτικά χωρισμένε έτσι ώστε αν θελήσουν να καθίσουν μαζί να πληρώσουν παραπάνω. Ενώ το μήνυμα είναι ότι απλά θα μπορέσουν να αλλάξουν τη θέση του. Ε, έχουν προκληθεί και διενέξει και με το πλήρωμα. Σε κάθε περίπτωση ε, μιλούμε για εκβιασμό, για προσπορισμό μεγαλύτερων κερδών από πλευρά τη Ryanair και άλλων τέτοιων ε, εταιριών. Αυτή η εταιρεία δημιουργεί εκ προημίου και εκ των προτέρων μια κατάσταση δυσχερή για να υποχρεώσει τους ε, επιβάτες να πληρώσουν αν θέλουν να ταξιδέψουν με, μη, με όχι τόσο δυσάρεστο τρόπο. Δημιουργείται στις συνθήκες δυσαρέσκειες για να υποχρεώσει την έξτρα χρέωση και την επιπρόσθετη ε, αγορά. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, έτσι ώστε να αλλάξουν συμπεριφορά οι εταιρείε χαμηλού κόστου και να φέρονται με πιο ανθρώπινο τρόπο στου επιβάτε του. Κυρία Πρόεδρε, εμεί οι καταναλωτέ, οι χρήσει, σα ζητούμε να υιοθετήσετε νομοθετικέ πρωτοβουλίε για να ρυθμιστεί ο τρόπο με τον οποίο πολλούνται αυτά τα εισιτήρια και έτσι ώστε οι εταιρείε που πετάνε στην Ευρώπη να ε, μην υποχρεώνουν αυτού που κάνουν ομοδικέ υποχρεωτική κράτηση να κάθονται χωριστά για να πληρώσουν έξτρα μετά. Να τους βάζουν μαζί, αφού μαζί θέλουν να ταξιδέψουν και μαζί αγοράζουν τα εισιτήρια και μαζί το δηλώνουν. Ε, να είναι κατά μέγιστο στην ίδια σειρά ε, ή τουλάχιστον στην αμέσω επόμενη. Ε, να υπάρξει νόμος γι' αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεσμευτική υποχρέωση να τους βάζω δίπλα-δίπλα ή τουλάχιστον στην ίδια σειρά ή σε δύο κοντινές σειρές. Θα πρέπει να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίτερ Σόρενσεν, παρακαλώ, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητέ κύριε Ροντρίγκεθ ε, Σάντσεθ, καλημέρα σε όλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα εμπορικό σκέλος και ένα σκέλος ασφαλείας σε σχέση με αυτή την αναφορά. Η απάντηση που έχουμε υποβάλει γραπτός και η απάντηση που θα δώσω σήμερα έχει να κάνει με την ασφάλεια. Δεν υπάρχουν νομικές ή ρυθμιστικές διατάξεις σε σχέση με τις εμπορικές ε, πρακτικές του να χρεώνει κανείς για να μοιράσει τις θέσεις. Το, η μόνη υποχρέωση του μεταφορέα είναι να το κάνει με διαφανή τρόπο, τον τρόπο με τον οποίο μοιράζει και δίδει τις θέσεις. Τώρα, από πλευρά ασφαλεία όμως, Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξει για τις αεροπορικέ μεταφορές, οι οποίες ε, έχουν καταγραφεί σε σχέση με τις θέσεις των ε, επιβατών. Και αυτό υπάρχει στην νομοθεσία 965 του 2012 για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις διοικητικές διαδικασίες για τις αερομεταφορές. Σε Καταρχάς, οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες ανάθεσης θέσης, έτσι ώστε οι επιβάτες να κάθονται με τρόπο ώστε η ασφάλεια εντός του αεροσκάφους να είναι σίγουρη να, και να μην υπάρχει ε, πρόσκομα στο ενδεχόμενο εκένωσης. Αυτές οι διατάξεις δεν είναι περιγραφικές γιατί είναι πολύ διαφορετικά τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται, ε, πολύ διαφορετικές υπηρεσίες που προσφέρονται. Λόγω της πλειάδας δηλαδή του αεροπορικού τοπίου δεν καταγράφονται ενδελεχώς αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες όμως πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να είναι καταγεγραμμένες και πρέπει να έχουν τύχη έγκριση στις Εθνικές Υπηρεσίες Πολιτικής ε, Αεροπορίας ούτω ώστε να μπορέσει η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία να εκδώσει πιστοποιητικό ότι μπορεί όχι μεταφορέ να πετάξει το αεροπλάνο του και έχουμε και κατηγορίες, ε, ειδικέ κατηγορίες επιβατών. Υπάρχουν διάφορες ειδικέ κατηγορίες ε, επιβατών, για παράδειγμα ε, επιβάτες με αναπηρίες, με προβλήματα όρασης ή ακοής και νομίζω ότι υπάρχουν και διατάξεις σε σχέση με τα ανήλικα τέκνα, με τα πολύ μικρά παιδιά με τα βρέφη κάτω των 24 μηνών, αλλά και με τα παιδιά ε, μικρής ηλικίας από 2 ως 12. Η αναφορά αυτή κάθε αυτή δεν αναφέρεται στην ευρύτερη περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων. Όμως, με το επιχειρήματα για τον ενδυνάμει διαχωρισμό των οικογενειών ως προς τη θέση που ε, θα καθίσουν, ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Υπ' αυτή την έννοια, στις διαδικασίες για το ποια θέση δίνουν στους επιβάτες οι αρωματαφορές αναφέρεται ότι ένα παιδί ειδική κατηγορίας επιβάτης δηλαδή, πρέπει να κάθεται δίπλα ε, στον ενήλικα που το συνοδεύει. Δηλαδή ε, το παιδί ε, εντάσσεται στην κατηγορία ειδικό επιβάτης που πρέπει να κάθεται μαζί με το συνοδό του. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει οι αερομεταφορείς να έχουν διατάξεις που, ε, να, έχουν διατάξεις που να, προβα... να επιτρέπουν έναν ελάχιστο διαχωρισμό. Δηλαδή, εάν πρέπει να χωριστούν αυτοί, πρέπει να χωριστούν το πολύ κατά μία σειρά ή κατά ένα διάδρομο. Η επικρατούσα αρχή είναι ότι όταν μεταφέρονται επιβάτες ειδική κατηγορίας θα πρέπει να μεταφέρονται υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια του αεροσκάφους και των επιβενόντων. Η ασφάλεια λοιπόν είναι ε, προτεραιότητα και επικρατεί έναντι των εμπορικών πρακτικών. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις εμπορικές πρακτικές τις επιχείρησης και του ρομεταφορέα, αλλά μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι διενεργούνται με ασφαλή τρόπο και για το ρεσκάφος και για την εταιρεία και για τους επιβαίνοντες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα. Έχουν το λόγο οι συνέλφοι της Επιτροπής μας. Εσείς, ε, συνάδελφοι, έχετε ζητήσει πρώτος το λόγο. Ο κύριος Αμέριξ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σάντζεθ, κατανοώ ότι θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση υπέρ των ε, επιβατών. Κυρίως για τις ε, οικογένειες. Όπως έχει σήμερα η καινοτική νομοθεσία υπάρχει ρύθμιση ενδελεχής. Είναι υποχρέωση της αεροπορικής εταιρεία να καλύψει τις ανάγκες ε, των οικογενειών και των ομάδων παιδιών που αναφέρατε. Πρέπει να, επίσης να υπάρχει πλαισίωση των παιδιών κατά από δύο έτη ηλικίας Επομένω υπάρχουν διάφορες διατάξει που ρυθμίζουν την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να νομοθετήσουμε περαιτέρω. Μας τα εξήγησε άλλωστε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασική μέρημνα βέβαια είναι η ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών. Τώρα όσον αφορά το να μπορούν να κάτσουν λοιπόν αυτοί οι επιβάτες που είπατε μαζί, ε, αυτό μπορεί να καλυφθεί με την ισχύωση νομοθεσία. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε την αναφορά η Πρόεδρος. Κύριε Σάντσα θα έχετε τον ε, λόγο για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντω ισχύει ένα κανισμό που μιλεί, μιλά για παιδιά ε, μικρότερα των δύο ετών που συνοδεύονται από τον γονέα τους. Αλλά έχουμε και το θέμα των ε, μη συνοδευομένων που είναι μέχρι 12 ετών. Επομένω, αυτό είναι διαφορετικό. Δεν μιλούμε για τους μη συνοδευόμενους, ούτε για τα μωρά αυτά, ε, γιατί αυτά όντως καλύπτονται από την νομοθεσία. Μιλούμε για οικογένειες που ταξιδεύουν με τα παιδιά τους που είναι 8 ή 10, είναι ανήλικοι και δεν είναι στέση να ταξιδέψουν με τους γονείς τους. Επομένως, δεν είναι θέμα άνεσης. Είναι θέμα ασφάλειας και όχι μόνο. Έχουμε και πρόσωπα με αναπηρία και οι αναπηρίες που δεν είναι ορατές. Δεν καλύπτονται αυτά. Φανταστείτε κάποιον που πάσχει σχιζοφρένεια ή κάποια άλλη αναπηρία που δεν είναι αισθητή ή ορατή και δεν, δεν, έχει, δεν μπορεί να κάτσει μαζί με την οικογένειά του. Ε, αυτό είναι θέμα ασφάλειας για όλους τους επιβάτες του αεροπλάνου. Και ο σκοπός μας είναι αυτός. Όχι η άνεση των υφατών, που φυσικά αυτό είναι θεμητό γιατί γι' αυτό πληρώνω. Αυτό που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα ασφάλειας. Γιατί αυτή η σύσταση τη κοινότητα του Κοινοβουλίου τέλο πάντων, επειδή δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, δεν τηρείται. Οπότε, είναι πολλά τα προβλήματα και αυτά τα προβλήματα μπορεί να είναι θέματα ασφαλείας. Παρακαλώ να το λάβετε αυτό υπόψη και να κρατήσετε ανοιχτή την αναφορά. Γιατί ενδεχομένως να έχουμε σοβαρά προβλήματα εάν συνεχίσουν αυτή την τακτική αεροπορικές εταιρείε ε, το κίνητρό του το μοναδικό του κίνητρο, το κέρδος. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ακούσαμε και τον Αναφέρονται εκτός από τους συναδέλφους και την Κομισιόν. Προτείνουμε να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Γιατί μα ανέφερε κάποιε εμπορικέ πρακτικέ η Επιτροπή που θα πρέπει να διέπονται και από τη μερική ασφάλεια αλλά και από διαφάνεια. Ακούσαμε τον αναφέροντα, ακούσαμε τους συναδέλφους και θα ζητήσουμε από την Επιτροπή των Μεταφορών να γνωμοδοτήσει, ούτω ώστε να αναβαθμιστεί η προστασία του καταναλωτή όσον αφορά αυτές τις εμπορικές πρακτικές. Ευχαριστούμε κύριε Ροντρίγκεθ. Να είστε βέβαιος. Εμείς έχουμε κατά νου τα συμφέροντα των καταναλωτών, των Ευρωπαίων. Για οποιαδήποτε αδικία και παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Πρόκειται για πολλές οικογένειες που ταξιδεύουν αεροπορικά, που σας ε, απασχόλησε το θέμα του. Πάμε τώρα στο σημείο 24 είναι η αναφορά 5 του 19 της Μπάρμπαρα Κλίμερ Γερμανίδας για ζητήματα μετανάστευσης στην Ελλάδα και ειδικότερα στο νησί της Σάμου. Δεν ήρθε η αναφέρουσα. Κύριε Κατερίνα Σταμάτη, έχει το λόγο από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Η αναφορά σχετίζεται με τον μεγάλο αριθμό μεταναστών που βρίσκονται στο νησί της Σάμου στην Ελλάδα και στις επιπτώσεις που αυτό έχει στη ζωή των ίδιων των μεταναστών αλλά και των ντόπιων κατοίκων στην αναφορά γίνεται έτοιμα για μετεγκατάσταση των ε, μεταναστών από την Ελλάδα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και για περισσότερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη πρωτοβουλειών υπέρ της με κάλυψη της μετανάστευσης. Το 2016 η Κομισιόν πρότεινε ένα νομοθετικό πακέτο για την μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου και περιλαμβάνει αυτό μία πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος του Δουβλίνου. Είναι οι κανόνες ε, που ορίζουν ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση μιας αίτησης ασύλου. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει έναν ε, διορθωμένο μηχανισμό μετεγκατάστασης, ο οποίος ε, θα διασφαλίσει ότι κανένα κράτος μέλος ε, δεν επιδέχεται δυσανάλογη πίεση και βάρος λόγω της μετανάστευσης. Όμως, επειδή αυτό ακόμα δεν έχει κριθεί από τους συνομοθέτες, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέχρι και η Κομισιόν βέβαια έχει επανειλημμένα αναφέρει την πλήρη αποφασιστικότητά της και τη δέσμευσή της ε, να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα και ότι αυτό πρέπει να κάνουν και τα κράτη-μέλη. Μέχρι λοιπόν να βρεθεί αυτή η συμφωνία, η Κομισιόν ενισχύει και υποστηρίζει τις ad hoc προσπάθειες των κρατών μελών να μετεγκαταστήσουν τον κόσμο. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, η χρηματοδότηση και υποστήριξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 και μετά να έρχεται σε πάνω από 2 δις ευρώ. Με αυτό το ποσό η Κομισιόν υποστήριξε τις ελληνικές αρχές σε πολλά επίπεδα της διαχείρισης της μετανάστευσης, όπως ας πούμε την στέγαση, την υποδοχή, διαδικασίας ασύλου, ιατρική βοήθεια, προστασία ανηλίκων και πολλά άλλα. Η Κομισιόν πάντοτε είναι έτοιμη να συνεχίσει να παράσχει οικονομική και άλλη μορφής βοήθεια στις ελληνικές αρχές όταν τις, τη χρειάζονται, ενώ ταυτόχρονα θυμίζει ότι οι ελληνικές αρχές είναι υπεύθυνε για την διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Κάποιος συνάδελφος θέλει το λόγο. Ο κύριος Αντέμοφ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα αντικαθιστώ τον κύριο Ράντεφ, τον συνάδελφο που δεν μπόρεσε να παραστεί και να σας αναπτύξει τη θέση της πολιτικής μας ομάδας. Το ΕΛΚ κατανοεί το ότι η κατάσταση στη ΣΑΜΟ είναι δύσκολη, διότι υπάρχουν και πολλοί μετανάστες. Ακούσαμε τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολουθεί τις εξελίξεις και προσφέρει οικονομική και τεχνική αρρωγή στην Ελλάδα. Ο αναφέρον θέλει η Ευρώπη να κάνει περισσότερα, να βοηθήσει περισσότερο σε σχέση με τις τοπικές μεταναστευτικές πρωτοβουλίες και να μην ε, επενδύει σε θέματα που δεν είναι προτεραιότητας. Φερρυπίν, μας αναφέρει εδώ τις επενδύσεις που έχουν γίνει για το τοπικό ναυτικό μουσείο. Αναφέρεται εδώ οι πρωτοβουλίε του Ταμείου τη Μετανάστευση. Ε, άλλο αυτό, αλλά και άλλο το θέμα του Ναυτικού Μουσείου. Δεν είναι δυνατόν να γίνει μεταφορά από οποιοδήποτε ταμείο σε ένα άλλο. Η νέα ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι πρόκειται να έχει καλύτερη στρατηγική όσον αφορά τους μετανάστες και ότι θα βελτιωθεί η κατάστασή τους στα νησιά και προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει κάποια μέτρα. Αυτό όμως χρειάζεται κάποιο χρόνο για να γίνει και θα οδηγήσει τελικά σε βελτίωση της κατάστασης. Θεωρούμε ότι πρέπει να κλείσει η αναφορά ως ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Nicolai Alavanos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τον συνάδελφο που πήρε το λόγο πριν. Κατά την άποψή μα είναι μια αναφορά η οποία πρέπει να μείνει ανοιχτή. Η αναφέρουσα περιγράφει μια εκρηκτική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες λόγω ακριβώς του διπλού εγκλωβισμού τους σε άθλιες συνθήκες στα hot spots της ΣΑΜΟΥ, αλλά και τις, δύσκολε δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες όχι μόνο στο νησί της ΣΑΜΟΥ, αλλά και στη Λέσβο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου. Από την κατάθεση της αναφοράς και από την απάντηση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής της προηγούμενης ελληνικής κυβέρνησης μέχρι και σήμερα έχει αλλάξει η κατάσταση. Βλέπουμε αύξηση των προσφυγικών, των προσφυγικών ροών, ιδιαίτερα μέσα στο καλοκαίρι, με συνέπεια την αύξηση των εγκλωβισμένων στα hot spots του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, στη Σάμο, σε δομέ που μπορούν να φιλοξενήσουν 700 με 800 άτομα, διαμένουν σε άθλιες συνθήκε πάνω, από 5.000. Στη Λέσβο είναι πάνω από 10.000 εκείνοι οι οποίοι διαμένουν σε δομέ που μπορούν να φιλοξενήσουν γύρω στου 1.000 με 1.500 ανθρώπου. Πρόκειται για hot spots φτιαγμένα με προδιαγραφέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο παραμένει, επομένω, η αιτία που δημιουργεί την προσφυγιά, τη μετανάστευση, που κατά την άποψή μα είναι ο πόλεμο, οι επεμβάσει, στι οποίε συμμετέχουν και κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα καμία λογική επαναπροώθηση, ούτε η καταστροφική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Κατά την άποψή μα, η μεταφορά στην ενδοχώρα από τα νησιά μερικών εκατοντάδων ε, ανθρώπων, όπως προτείνει η νέα κυβέρνηση, ή η οικογενειακή επανένωση μόνο μερικών ανηλίκων, δεν λύνει το πρόβλημα. Όσο παραμένουν σε ισχύ οι περιορισμοί που βάζει, για παράδειγμα, ο κανονισμός του Δουβλίνου, βλέπουμε στη δημοσιότητα να, έρχεται, να έρχονται στοιχεία του νέου σχεδίου για το Δουβλίνο 4, το οποίο είναι ακόμα αρνητικότερο, μιλάει ακόμη και για κανόνες εμπλοκής, όσο παραμένουν, ε, όσο αυξάνεται η εμπλοκή της Frontex και του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, που δεν λύνει το πρόβλημα, όσο σκληραίνει η ελληνική κυβέρνηση με βάση τι ανακοινώσει τη, τι διαδικασίε χορήγησης του ασύλου, για παράδειγμα με την πρόταση για την κατάργηση τη δευτεροβάθμιας εξέταση των αιτήσεων. Κατά την άποψή μα, αυτό που χρειάζεται να υποστηριχθεί σε αυτή τη φάση είναι ότι πρέπει να κλείσουν τα hot spots, αυτέ οι άθλιε δομέ που υπάρχουν, να μεταφερθούν οι πρόσφυγε και οι μετανάστες σε αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενία τη υπηρετική Ελλάδα, όπου εκεί θα εξετάζονται τα αιτήματά του και στη συνέχεια θα πηγαίνουν στι χώρε πραγματικού προορισμού, να προχωρήσουν άμεσα οι, οικογενο... οι οικογενειακές επανενώσεις έτσι ώστε κανένα ανήλικο, να μην ζει σε ακατάλληλες συνθήκε, να μην ζει απροστάτευτο, να μην ζει άστεγος ή φυλακισμένο, και βεβαίω να παρθούν μέτρα έτσι ώστε να αποζημιωθούν στο 100% οι νησιώτες οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές από το διπλό εγκλωβισμό που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο κύριος Άκους Σαλμπία. Είμαι πολίτης από μια χώρα που είναι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Μάλτα, και καταλαβαίνω και καταναώ πλήρως την αναφέρουσα. Ε, η αλληλεγγύη δεν φαίνεται στην Ευρώπη σε θέματα μετανάστευσης και πολύ σωστά ζητάει κανείς την αλληλεγγύη. Μα σταμάτησαν από το να μιλάμε για την αναθεώρηση του Δουβλίνου εδώ και τέσσερα χρόνια. Τραγωδίες σημειώνονται στις θάλασσές μας και πρέπει όλα τα κρατημέλη να αναλάβουν σοβαρή δράση. Πρέπει να δοθεί περισσότερη βοήθεια στα κράτη-μέλη που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης για να σταματήσουν αυτές οι ανθρώπινες τραγωδίες. Ε, απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να διατηρήσει την αναφορά ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχοντας διαβάσει την αναφορά, έχοντας ακούσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας ακούσει τα μέλη της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναφορών, προτείνω ως Πρόεδρος να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή. Θα στείλουμε, στείλαμε στις 3 Ιουνίου τη σχετική πληροφόρηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση στα ελληνικά νησιά, δίνει τεχνική και οικονομική βοήθεια στις ε, εθνικές αρχές για να απαλληθεί η φυστάμενη μεταναστευτική πίεση. Έχει προτείνει νομοθετικό πακέτο για την αναθεώρηση του Δουβλίνου που θα πρέπει να εγκριθεί από τους συνομοθέτες. Υπάρχει νέα επιτροπή, θα υπάρξουν νέοι επίτροποι. Επομένως, εν ώψη όλων αυτών πρέπει η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή έτσι ώστε η επιτροπή να μας ενημερώσει ε, για το νομοθετικό πακέτο, την νομοθετική δέσμη μέτρων που παραμένει εκρεμής και θα πρέπει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να μας ενημερώσει για τη συμβατότητα με την ε, κοινοτική νομοθεσία και για το κατά πόσο τηρούνται τα δέοντα. Αυτά προτείνει η Προεδρία λοιπόν της Επιτροπής σας. Περνάμε στην αναφορά 0695-2017, σημείο 25 της ημερήσιας διάταξης, αναφορά που υποβλήθηκε από Ιταλό πολίτη για την αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και την πρόσβαση των αστέγων πολιτών σε υγειονομική περίθαλψη. Η αναφέρουσα δεν είναι παρούσα και γι' αυτό θα θέλαμε να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία ε, Ζωζεφίνα Χάδερστρομ. Ε, thank you, Madam eh, ε, Αγαπητέ Πρόεδρε της Επιτροπής, να δώσω μια γενική δήλωση για τις κοινωνικές πολιτικές ε, έχουν συμβεί πολλά από τότε που έγινε, δόθηκε αυτή η απάντηση. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η έλλειψη στέγης είναι μια ακραία κατάσταση και έχει διαπιστώσει την αύξηση της έλλειψης στέγης σε διάφορα κράτη-μέλη πέραν της Φιλανδίας. Το να βελτιώσουμε ε, τι στεγαστικές συνθήκες των ευάλωτων ομάδων και η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ε, για αυτά τα θέματα είναι μέσα στις 20 βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Να θυμίσω ότι η συνθήκη δεν δίνει την εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ε, προγράμματα κοινωνικής αρρωγής στα κράτη-μέλη. Αυτές είναι αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της συνθήκης, η Επιτροπή συμπληρώνει τις δράσεις και υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στη μάχη τους κατά ε, της έλλειψης στέγης και των αποκλεισμών. Η Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή 19 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για τη στέγαση και την βοήθεια στους αστέγους. Επίσης, έχει μια πολιτική καθοδήγηση ε, ε, τη χρήση κοινωνικών ε, ταμείων όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ε, το Ταμείο για την Ανέχεια, για την ακραία φτώχεια. Αυτά είναι χρηματοδότηση από την Κομισιόν και η Κομισιόν παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών στο θέμα της έλλειψης στέγης και των αποκλεισμών. Από την τελευταία απάντηση της Κομισιόν έχει ε, αλλάξει το γεγονός ότι ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων έχει ε, ανακηρυχθεί από τα κράτη-μέλη ως ένας βασικός πυλώνας ε, και ε, υπάρχει η αρχή 19 που τον διέπει. Ε, φαίνεται ότι στις διάφορες ε, εκθέσεις για τις χώρες που γινόνται μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αναφέρεται η έλλειψη στέγης και στάλησαν ήδη οδηγίες για τη βελτίωση και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς στέγασης. Υπάρχει περισσότερη έμφαση στη στέγαση των ευάλωτων ομάδων. Φέτος πολλές χώρες πήραν συστάσεις, υπάρχουν 8 κράτη-μέλη. Τα τέσσερα ε, έχουν ε, δεχτεί συστάσεις σχετικά με τις επενδύσεις. Επίσης, η Κομισιόν συνεχίζει να προωθεί τη συζήτηση, ε, την ανταλλαγή μαθημάτων και πρακτικών για την αντιμετώπιση των αποκλεισμών και της έλλειψης στέγης. Υπάρχουν συναντήσεις που γίνονται μέσα και υπό την αιγίδα της Φιλανδικής Προεδρίας, για παράδειγμα. Επιπλέον, στο μέλλον η Κομισιόν θα συνεχίσει να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την πρόσβαση των πολιτών στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Κομισιόν θα θέσει τις προτεραιότητες, θα δώσει τα εργαλεία που θα βοηθήσουν προς αυτό το στόχο. Να καταλήξω και με δύο ε, σχόλια για την πρόσβαση στα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Χάρτα για τα θεμελιώδη δικαιώματα αναγνωρίζει στο άρθρο 14 το δικαίωμα για τη στέγαση και για τη βοήθηση. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επίσης μίλησε για το δικαίωμα της ε, ιδιωτικότητας υπό το άρθρο 7. Η χάρτα ε, εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης αναγνωρίζει το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών, το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε στις ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές ε, ως ε, ε, κανονικοί πολίτες της κάθε χώρας. Δεν έχει γενική εξουσία να παρεμβαίνει σε εθνικά βέβαια, εκλογικά θέματα η Κομισιόν. Η εφαρμογή του Εθνικού Εκλογικού Νόμου υπόκειται στη δικαιοδοσία των αρχών των κρατών μελών. Για να διευκολυνθεί όμως η φυσιολογική συμμετοχή των ανθρώπων που ε, απειλούνται με αποκλεισμό στην τοπική τους κοινωνία, ε, έχει ε, θεσπιστεί η δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν έναν λογαριασμό με κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Στην Ιταλία έχουμε λογαριασμούς πληρωμών που έχουν βασικά χαρακτηριστικά και απευθύνεται σε συνταξιούχους και άλλους ε, τέτοιους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι η σειρά των μελών της Επιτροπής. Η κυρία Ντανόκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κρίμα που δεν έχουμε τους αναφέροντες παρόντες. Την αναφέρουσα. Είναι όμως ενδιαφέρουσα αναφορά αυτή. Είναι μη ικανοποιητική η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αναφέρουσα είναι άστεγη. Αλλά μιλάει για τα εργασιακά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα με την ιδιότητά του του άστεγου πολίτη. Ναι, αγωνιζόμαστε ενάντια στη φτώχεια, την ακραία φτώχεια. και το φαινόμενο των άστεγων πολιτών. Όμως δεν απεκδίονται οι άνθρωποι τα δικαιώματά τους βάσει του κώδικα πολιτικής δικαιονομίας, βάσει του νόμου, επειδή είναι άστεγοι. Είναι πρόβλημα το να λάβει ταυτότητα, το τονίζει αυτό η αναφέρουσα, το οποίο είναι το βασικό έγγραφο, που της επιτρέπει να είναι ενεργός και πολιτικός δραστήρια. Πρότασή μου λοιπόν είναι να το μελετήσουμε αυτό το θέμα και να κάνουμε μια καταγραφή πώς στα διάφορα κράτη-μέλη αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν ε, σπίτι, σταθερή κατοικία. Και κατά πόσο δυσκολεύονται να ασκήσουν ε, βασικά δικαιώματά τους που απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη. Στη χώρα μου, Στη χώρα μου, ε, για παράδειγμα, για να συμμετάσχει κάποιο σε ευρωεκλογέ, αν είναι ξένο, ναι, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει τη διεύθυνσή του για να γνωρίζουμε ότι όντω ζει εδώ και άρα δικαιούται να συμμετάσχει σε εκλογέ. Αυτό είναι λογικό. Αλλά γιατί να χρειάζεται για τους αστέγους πολίτες. Ε, χρειάζεται απλά μια πιστοποίηση ότι ζουν, ότι είναι πολίτες και ότι μπορούν κάλλιστα να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για τους ξένους που θέλουν να συμμετάσχουν στις δημοτικές τοπικές εκλογές. Γιατί δηλαδή ε, το να μην δύναται κανείς να προσκομίσει διεύθυνση να είναι λόγος για να αποκλείεται από ορισμένα δικαιώματά του. Πρέπει να μελετηθεί αυτό το θέμα, ίσως αποκοινούμε την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντιπρόεδρε. Από πλευράς ΕΛΚΑ, παρακαλώ, το λόγο έχει ο κύριος Βίντσε. Ευχαριστούμε τον ε, αναφέροντα. Ήταν πολύ δύσκολο γίνουν. Ε, ακόμα και η μετάβασή του στις Βρυξέλλες ήταν ένα ζήτημα. Ε, Βεβαίω και ακριβώς αυτό αφορά η αναφορά του. Γιατί ε, είναι μια προσωπική τραγωδία η υπόθεση των ε, αστέγων. Πάντα υπάρχει μια τραγωδία πίσω από την ε, προσωπική ιστορία του κάθε άστεγου. Θεωρώ ότι τα δικαιώματα αυτών των πολιτών δεν ισχύουν, μια που δεν έχουν επίσημη διεύθυνση, δεν έχουν επίσημα έγγραφα και επομένω ε, δεν μπορούν να έχουν κάποιε κοινοφελεί υπηρεσίε, δεν μπορούν να ασκήσουν τα πολιτικά του δικαιώματα. Δεν έχουν πρόσβαση στι κοινωνικέ, υγειονομικέ υπηρεσίε, δεν μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό κλπ. Νομίζω ότι θα πρέπει να εκπαινέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειές της. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για φαινόμενο το οποίο τώρα εξελίσσεται. Θα πρέπει ε, τα κρατημέλη να το λάβουν υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δέσμη ελαχίστων δικαιωμάτων για τους αστέγους να είναι καταγεγραμμένοι σε κάποιο μητρό. Έτσι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κάποια αγαθά και κάποιες υπηρεσίες, όπως Φερρυπίν, το να μπορούν να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό. Βέβαια, είναι θέμα κοινωνικό, είναι θέμα οικονομικό. Ε, το πρόβλημα του δεν έχουν στέγη. Όσον αφορά τώρα την συγκεκριμένη αναφορά, θεωρώ ότι θα πρέπει να κλείσει. Όμως, θα πρέπει η προβληματική να συνεχιστεί. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε κάποιες ε, ενδελεχείς συστάσεις προς τα κάτι μέλη. Κάθε περίπτωση φυσικά είναι διαφορετική, αλλά χρειάζεται η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τώρα να καταβληθούν προσπάθειες από την Ευρώπη. Αυτό θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις θέσεις των συναδέλφων και τις θέσεις του αναφέροντος. Είναι εθνική αρμοδιότητα, ακούσαμε και για συγκεκριμένες, ε, ε, υποθέσεις του αναφέροντος δεν μπορεί να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται όμως για σοβαρό θέμα για το ότι κάποιος δεν έχει δικαίωμα σε στέγαση και στην Ιταλία και σε άλλα κράτη-μέλη. Ε, είχαμε και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ε, είχαμε τον κοινωνικό πυλώνα για τα θέματα κοινωνικού αποκλεισμού. Οπότε, Περιμένω την έκθεση του 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε πρόκειται να δημοσιοποιηθούν τα σχετικά στοιχεία για τους άστεγους, για τον ε, αποκλεισμό, για την γεωργική πολιτική σχετικά με αυτά του κάθε κράτους μέλους. Οπότε την ε, αναφορά κατευθείαν την κλείσουμε. Αλλά όλες τις πολιτικές ομάδες, όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει ε, σύμφωνα με την προθεσμία που είπαμε χτες τα είπαμε στους συντονιστές, θα πρέπει μέσα αυτή την προθεσμία να ζητήσουμε η λίμπε να κάνει όλα αυτά τα οποία μας ενέφερε και η κυρία Ντάνοκα και ο κύριος Βίντζε. Αυτά σας προτείνω. Και τώρα, προχωρούμε στην επόμενη αναφορά που είναι το σημείο 26. Πρόκειται για την αναφορά 535 του 2017 που την έχει υποβάλει ο κύριος Λουντό Έρμαντς που είναι Βέλγος και αφορά τις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε, κύριε, πέντε λεπτά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Πάντοτε ακούμε προσοχή τους ε, Ευρωπαίους. Πέντε λεπτά. Δεν ακούγεστε. Α, ε, Δεν έχετε ανάψει το μικρόφωνο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ που μελετάτε την αναφορά μου. Σας την υπέβαλα σε εσά, αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε κάποια παρεξήγηση Συγγνώμη φορώ το καπέλο γιατί έχω προβλήματα όρασης που το προκαλεί το φως. Άλλα ισχύουν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα όσον αφορά τους ανθρώπους με αναπηρία και επίσης αυτές τις ειδικέ κάρτες που δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ε, σε κάποιες εκδηλώσεις ε, κοινωνικές και πολιτιστικές. Αυτό το πάσο, ας το πούμε. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Κράτη Αναπηρίας, αλλά δεν σχετίζεται με τα θέματα μετακίνησης. Μετακίνησης των ανθρώπων με αναπηρία. Οκτώ χώρες μόνο συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση, όπως σας τα είπα και στο έγγραφο. Είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένη χώρα η κάρτα. Οπότε άπαξ και κανείς περάσει τα σύνορα της χώρας του δεν μπορεί να έχει τέτοια κάρτα. Πάντως το βασικό θέμα είναι η μετακίνηση, η κινητικότητα που λέμε, το με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αναπηρία δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη χώρα. Είναι προσωποπαγές ζήτημα. Δεν σταματά το πρόβλημα στα σύνορα, οπότε αν κάνει έχει κάποιο πάσο σχετικό, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε κάποια άλλη χώρα. Αν λοιπόν θέλει να πάει σε άλλη χώρα κάποιο με αναπηρία θα πρέπει για τον σύνοδο, τον οδηγό του τέλο πάντων να πληρώσει επιπλέον. Αυτό είναι κάποιο είδου διάκριση. Γιατί ο οικονομισμό προβλέπει ότι άνθρωποι με αναπηρία ε, δεν μπορεί να τους απογραφεί η πρόσβαση κάπου ε, και βέβαια αυτό αφορά τις τα μαξίδια τέλος πάντων. Αλλά ε, συστήνει ο κανονισμός ότι θα πρέπει κάποιες ώρες πριν να ανακοινώσει το ότι μετακινείται. Το e-links αυτό αφορά τέσσερις χώρες τις οποίες είναι υποχρεωτική η ειδοποίηση. Άρα δεν είναι ελεύθερη η διακίνηση των ανθρώπων με αναπηρία ε, αυτών των ανθρώπων που έχουν ανάγκη οδηγού, συνοδού. Οπότε μετά είναι το θέμα ότι ο οδηγό θα είναι από άλλη χώρα κλπ. Αυτό που ζητούμε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα αναγνωρίζεται από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες η αναπηρία κάποιου που προέρχεται από κάποια χώρα μέλος και αντιστοίχως θα πρέπει να είναι έγκυρα τα πάσα αυτή και οι κάρτες από οποιαδήποτε χώρα. Οπότε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς επιπλέον έξοδα να συμμετάσχουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και πολιτιστικέ ε, εκδηλώσεις. Περιμένω τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ελπίζω ότι θα υπάρξει αυτή η σωστή αντιμετώπιση των ανθρώπων με αναπηρία. Άρα αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να εξασφαλίσει ότι οι ανάπηροι που έχουν αυτό το πάσο θα μπορούν να ε, ταξιδέψουν, να διακινηθούν χωρίς επιπλέον έξοδα. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζωζεφίν Θα βγω για, για τρία λεπτάκια και δίνω τη σκητάλη στην αντιπρόεδρο Ντανόκα. Ευχαριστώ τον αναφέροντα, ευχαριστώ την κυρία Πρόεδρο. Θα χωρίσω την απάντησή μου σε δύο ε, τμήματα. Πρώτα μια γενική δήλωση και μετά ενημέρωση για το τι κάνει η Κομισιόν από την τελευταία της απάντηση και μετά. Η Επιτροπή αναγνωρίζει τις προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία καθώς ταξιδεύουν στα κράτη-μέλη, ειδικά όταν ε, το καθεστώς της αναπηρίας και οι εθνικές κάρτες αναπηρίας δεν αναγνωρίζονται από κάποιο κράτος μέλος. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε πιλωτικά το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας σε 8 χώρες. Είναι ένα θελούσιο σύστημα το οποίο ε, ε, αφορά στην αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασης της αναπηρίας μεταξύ των κρατών μελών. Τα κράτη εθελοντικά ε, παρέχουν τις ε, ίδιες ε, παροχές ε, όπως ας πούμε στο τομέα του πολιτισμού, της μεταφοράς, του αθλητισμού. Εκεί θα δούμε αν θα περιληφθούν συγκεκριμένες παροχές σε αυτό το project. Γενικά, οι διάφορες χώρες έκαναν η κάθε μία τη δική τους επιλογή. Όσον αφορά τώρα τους προσωπικούς βοηθούς, δεν έχουν όλοι συμφωνήσει να παρέχονται δωρεάν, ούτε περιλαμβάνουν στο σύστημά τους αυτή την ε, ε, ε, διευκόλυνση. Παρόλο που όλα περιλαμβάνουν τις μεταφο... και δεν περιλαμβάνουν και όλα τις μεταφορές. Επίσης, χρειάζεται αμοιβαία αναγνώριση για να βοηθούν τα άτομα με αναπηρία. Πρέπει η κατάσταση της αναπηρίας να πούμε ότι είναι στη δικαιοδοσία του κράτους ε, δεν υπάρχει εναρμόνιση των παροχών, άρα απάντοτε εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, το project της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, ε, τουλάχιστον σε λίγους τομείς, ε, βοηθά και ευαισθητοποιεί τους ενδιαφερόμενους στα αντίστοιχα κράτη-μέλη. Το δεύτερο κομμάτι είναι τι κάνουμε τώρα. Τώρα αυτή, αξιολογούμε αυτά τα, αυτή τη project εθελοντικής συμμετοχής που θα ολοκληρωθούν το 2020. Υπάρχει ένας εξωτερικός συνεργάτης, ένας ανάδοχος που ε, μπλέκεται σε αυτό και θα μας δώσει πληροφορίες. Επίσης, έχουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία για το 2020 όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγησή της, η Κομισιόν θα αποφασίσει τα μέτρα που θα προτείνει στο μέλλον σε, αυτόν τον τομέα. Επίσης, τα μέρη, ε, και άλλα κράτη-μέλη μπορούν να μπουν και αυτά στο πρόγραμμα με δικά τους ε, έξοδα, με δικές τους δαπάνες. Επίσης, η Κομισιόν εργάζεται συστηματικά για την άρση των φραγμών στη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρία σε δραστηριότητες όπως για παράδειγμα τα ταξίδια και οι μεταφορές. Έχουμε τους κανονισμούς για τα δικαιώματα των επιβατών. Έχω το συνάλφο εδώ που θα μπορούσε να δώσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες για αυτό το θέμα. Επίσης υπάρχει πρόσφατα η έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράξης για την προσβασιμότητα προσβασιμότητα σε μεγάλη γκάμα τομέων γιατί από ό,τι φαίνεται η προσβασιμότητα αυτή καθεαυτή μπορεί να διευκολύνει την ανεξαρτητοποίηση και την ε, ανεξάρτητη διαβίωση των ανθρώπων αυτών που πάσχουν από αναπηρία. Παρακαλώ, ο συνάδελφός σας θα ήθελε να προσθέσει κάποια στοιχεία από ό,τι κατάλαβα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας ε, στις δημόσιες μεταφορές και γενικότερα στις μεταφορές, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κανονισμούς για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλες τις μορφές ε, μεταφορών, ε, οδικές, ε, λεωφορεία, αεροπορικές, άλτομα με μειωμένη κινητικότητα. Πρέπει πάντοτε να μεταφέρονται, να μην τους αρνείται η επιβίβαση, να μην τους αρνούνται την επιβίβαση, να μην πληρώνουν επιπλέον εισιτήριο και να έχουν δωρεάν υποστήριξη και βοήθεια. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που να ορίζουν ποιο είναι το άτομο με μειωμένη κινητικότητα. Περιλαμβάνει ορισμός μια σειρά ατόμων. Οι κανόνες αυτοί βασικά θεωρούν ότι το ίδιο το άτομο πρέπει να δηλώσει ότι είναι άτομο με μειωμένη κινητικότητα. Ας πούμε, μπορεί να σπάσεις το πόδι σου και να έχεις γύψο. Μπορεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα να είσαι άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Άρα η εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί σε έναν τέτοιο επιβάτη την επιβίβαση, αλλά και πρέπει να του παράσχει και βοήθεια δωρεάν. Κύριε Χέρμανς, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κρατημέλη και κάποιοι μεταφορείς που μεταφέρουν και έναν βοηθό που συνοδεύει το άτομο χωρίς επιπλέον κόστος. Όμως δεν υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, κυρίως εξαρτάται από τα κράτη-μέλη και από τον μεταφορέα το πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα. Αυτό που λέω εγώ ε, ε, είναι ότι στις οδικές μεταφορές, με λεωφορεία, πούλμαν και στις πλωτές μεταφορές, ένα άτομο μπορεί να μεταφερθεί με βοηθό μόνο και όταν ταξιδεύει μόνο του, και δεν μπορεί να μεταφερθεί τελικά άμα δεν έχει βοηθό, θα πρέπει να μεταφέρεται μαζί του δωρεάν και ο βοηθός. Ε, στις σιδηροδρομικές και αεροπορικές μεταφορές δεν υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις. Για τις αεροπορικές ε, υπάρχει μια σύσταση στις ε, εταιρείε ε, να μεταφέρουν δωρεάν τους βοηθούς ή τουλάχιστον με μειωμένη τιμή. Νομίζω ότι αυτό θα ήθελα μόνο να προσθέσω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο και στον εαυτό μου, αφού... Γιατί και εγώ είχα, Γιατί εγώ είχα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το νομοθέτημα στην Επιτροπή Απασχόλησης. Και δυστυχώς ο νόμος για την προσβασιμότητα δεν προβλέπει διατάξεις για τη συνοδεία άλλων ατόμων διαφορετικών από το άτομο με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα αυτό καθ' αυτό. Επομένως, ο νόμος αυτός δεν έχει σχέση με την αναφορά σας γιατί το πρόβλημά σας είναι για τα δικαιώματα των συνοδών των ατόμων με αναπηρία. Ευχαριστούμε την Επιτροπή που εργάζεται πάνω, από αυτό, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν έχουν ληφθεί απαντήσεις από όλα τα κράτη-μέλη για το ζήτημα αυτό. Θα συνεχιστεί λοιπόν η εξέταση. Προτείνω. Ή να ακούσουμε και τον αναφέροντα. Από τα μέλη. Ναι. Κανείς δεν ζήτησε το λόγο. Δεν σας είχα δει, κύριε Άγγιου Σαλίμπια. Παρακαλώ, τοποθετηθείτε για την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι δύσκολη πρόκληση για ένα άτομο με αναπηρία να διάγει τον καθημερινό του βίο. δεν θα πρέπει να του περιπλέκεται η κατάσταση όταν επιλέγει να διαταξιδέψει στο εξωτερικό. Ε, λείπει εναρμόνιση και το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αυτό είναι σαφέστατα, σαφές. Αλλά θέλω να ασχοληθώ με τις κατευθυντήρες γραμμές για την ε, ε, κοινοποίηση των ε, που έχει καταγράψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν άρθρα που διατυπώνουν ξεκάθαρα ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να ζουν ανεξάρτητα και να ε, συμμετέχουν σε όλες τις πτυχές της ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει αυτή τη σύμβαση του ΟΗΕ και οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να έχουν ίση πρόσβαση ε, στο δικαίωμα των μεταφορών. Είχαμε το 2012 το έγγραφο εργασία για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλά ε, για μια ε, πρώτερη γνωστοποίηση 38 ώρων που πρέπει να δίδεται 48 ώρων για να, ότι θα ταξιδέψει άτομο με αναπηρία για να μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες αναδιατάξεις. Νομίζω ότι αυτή η προθεσμία των 48 ωρών για μεταφορά εναέρια, χερσαία ή θαλάσσια και η άλλη προθεσμία για τις οδικές μεταφορές, όλα αυτά είναι απαξιωμένα, είναι, ανήκουν στο παρελθόν. Πρέπει οι αεροπορικέ εταιρείε και οι άλλε να αξιοποιήσουν ε, τη νέα τεχνολογία, την οποία χρησιμοποιούν και τα άτομα με αναπηρίε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άτομα με μειωμένη κινητικότητα θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε όλου του τρόπου μεταφορά, όπω κάθε ένα από του υπόλοιπου πολίτε. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην κλείσει αυτή την αναφορά. Αυτέ οι χρονικέ ε, προθεσμίε είναι τεράστιες, είναι τελείω απαξιωμένε και απειρχαιωμένε ε, και αντιβαίνουν, αντίκειται στα δικαιώματα των ατόμων. Ευχαριστώ κύριο Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τον αναφέροντα και τους εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η αναφορά που συζητούμε γιατί έχει να κάνει με τα δικαιώματα περίπου 80 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών με διάφορα είδη αναπηριών. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν κυρώσει τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, αυτή η ομάδα πολιτών μας, συμπολιτών μας, αντιμετωπίζει, ε, προσκρούει σε εμπόδια που καθιστούν δυσχερή την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους. Και ένα από τα βασικότερα μελήματα και καθήκοντα του Κοινοβουλίου μας είναι να καταρρύψει αυτά τα εμπόδια και να εξαλείψει κάθε είδους ε, διακρίσεις. Ο κ. Χαϊμάς μας έχει ε, αναδείξει επανειλημμένος ότι όλα αυτά οφείλονται στο ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο έγγραφο που να έχει ε, γίνει να έχει εγκριθεί από όλα τα κρατη που θα επιβεβαιώνει ότι το εν λόγω άτομο έχει αναπηρία και άρα αυτομάτως είναι δικαιούχος ε, ε, είναι δικαιούχος για ε, να υπάρξουν οι σωστές ε, διατάξεις και ρυθμίσεις έτσι ώστε να έχει ίση πρόσβαση και έτσι θα μπορούσε να έχει μια ευρωπαϊκή κάρτα ε, ατόμου με αναπηρία για να αναγνωρίζεται παντού το καθεστώς του. η, πολιτική, η πιλωτική δράση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, καλή και καλούμε όλα τα κρατημέλη να θεσπίσουν νομοθεσία για να υιοθετήσουν αυτό το έγγραφο περιμένουμε με αγωνία και αδημονία να λάβει τις τελικές του πιναλιές αυτό το πολύ σημαντικό έγγραφο, το οποίο θα βοηθήσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους, θα βελτιώσει την πρόσβασή τους σε ισότιμη βάση στο χώρο εργασίας, στα πολιτιστικά αγαθά, στην εκπαίδευση, ε, στα ταξίδια, στην μετακίνηση εντός και εκτός των εθνικών συνόρων. Υπάρχει και το θέμα των επιβατών με αναπηρίες, το δικαίωμα δηλαδή της βοήθειας, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ε, να προειδοποιήσει εκ των προτέρων για την βούλησή του να ταξιδέψει με τόσο μεγάλη χρονική προθεσμία. Εμείς στο Κοινοβούλιο υιοθετήσαμε μια έκθεση πολύ φιλόδοξη για τους επιβάτες των σιδηροδρομικών μεταφορών όπου εξαλείψαμε αυτό το προαπαιτούμενο να έχει ενημερώσει εκ των προτέρων και μάλιστα 48 ώρες πριν ότι πρόκειται για άτομο με αναπηρία. Πιστεύουμε ότι η Φιλανδική Προεδρία θα οριστικοποιήσει ε, τη δουλειά για αυτό το τόσο σημαντικό έγγραφο. Νομίζω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η τελική εκδοχή του εγγράφου ταιριάζει και προσαρμόζεται σωστά στις ανάγκες των επιβατών μας με αναπηρίες. Και ελπίζω ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να λέμε ότι οι νέοι κανόνες, οι νέες λύσεις που έχουν υιοθετηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Ανάγκες οι οποίες σαφέστατα ανέδειξε ο κύριος Χέρμαν με την αναφορά του και τον ευχαριστώ για την πράξη του αυτή. Εκ μέρους του ΕΛΚ θα ήθελα η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο αναφέρον για δύο λεπτά παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας. Πρέπει να ε, πιέσετε το, το, να ανοίξετε το μικρόφωνο. Έχετε δύο λεπτά ακόμα θέλει για να κλείσετε την ε, αναφορά. Άκουσα τους βουλευτές και κατόπιν αυτό που άκουσα θεωρώ ότι δεν κλείνει, ότι παραμένει ανοιχτή η αναφορά και συνεχίζεται τις προσπάθειες για να δοθεί αυτή η δυνατότητα στους ανθρώπους με αναπηρία να μπορούν ελεύθερα να ταξιδεύουν παντού χωρίς φραγμούς και επιπλέον έξοδα για κάποιο σύνοδο. Ακριβώς όπως γίνεται και σε κάποιες μη ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε τελώ ένα αναμονή. Το 2013 έκανε τις πρώτες προσπάθειες και μου είπανε περίμενε, περίμενε και ακόμα περιμένω. Οπότε ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει κάποια βήματα πρόοδου και θα κάνει κάτι όπως προβλέπει το σχετικό κείμενο του ΟΗΕ, ούτως ώστε να είναι δυνατόν κάποιο να συνοδεύσει τον, συγγνώμη, να ταξιδέψει με τον συνοδό του χωρίς επιπλέον έξοδα, ε, ε, έξοδο, ούτως ώστε να μπορεί να συμμετέχει στα πολιτιστικά και δεν μιλώ μόνο για τη χώρα του ενδιαφερομένου, αλλά να μπορεί να πάει και σε άλλες χώρες, να περάσει τα σύνορα. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ακούσαμε τον αναφέροντα, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τους συναδέλφους, μέλη της Επιτροπής. Οπότε θα κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά. Έχουμε στείλει για ενημέρωση στην Τράνη, στην Ίμκο, και στην Επιτροπή Απασχόληση. το, Νοέμβριο του 2017 έγιναν όλα αυτά που ήρθατε στην συνεδρίασή μας στη συνέχεια τον Απρίλιο του 2018 και αποφασίστηκε να υποβληθεί η ε, αναφορά Ε, στους αρμοδίους και στους αρμοδίους ε, της περιφέρειας των Ευρωπαϊκών, αλλά ακόμα από η Γερμανία, η Ιταλία, Κύπρο και κάτω χώρες ε, επίσης αναμένουμε ενέργειες. Οπότε σας προτείνουμε να μην είναι ανοιχτή αναφορά. Οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη που δεν έχουν απαντήσει θα πρέπει να απαντήσουν ε, κατόπιν της επιστολής που θα τους ε, στείλουμε και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ενημερώσει κατόπιν ε, των νέων στοιχείων να στείλουμε, είπαμε, τα στοιχεία στην Επιτροπή Επασχόλησης για ενημέρωση, αλλά και στο Intergroup για τους ανθρώπου με αναπηρία, αλλά και στο European Framework, όπως προβλέπει το άρθρο 33. Μας στον, ε, στην Επιτροπή για Δημιουργία Δικαιώματα, στον Δημοσιολαβητή ε, και σε άλλο συναρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Οπότε θα υπάρξει παρακολούθηση εξέλιξη αναφορά σα και θα μείνει ανοιχτή. Και ευχαριστούμε πάλι που ήρθατε. Τελειώσαμε. Η επόμενη συνεδρίασή μα είναι 2 και 3 Οκτωβρίου. Τότε θα τα ξαναπούμε εδώ στις Βρυξέλλες. Γεια σας.